Colleagues, sorry. We are not very strong here. Είμαστε και τόσο πολλοί, αλλά είμαστε οι καλύτεροι. two from concern of... Αλλά οι σοσιαλιστές είναι οι καλύτεροι. Να το γεγονός ότι είναι δύο της GUE εδώ με ανησυχεί κάπως. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε πληροφόρηση για δύο σημαντικές συναντήσεις κορυφής Ιαπωνία. Θα αρχίσουμε διαπραγματεύσει για εταιρική σχέση συμφωνίας ε, και για συμφωνία ελεύθερο και με την Κίνα. Και έχουμε εδώ τον κύριο Ντέβιντο Σάλιμα και του δίνουμε το λόγο. Α κάνουμε και τα δύο θέματα μαζί, γιατί υπάρχει συνάθεια μεταξύ τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ε, που απασχοληθήκαμε πολύ με την Ασία αυτό το μήνα. Αρχές Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με την Κορέα, συνεχεία με, την... με τις συνόδους κορυφής ε, την περασμένη εβδομάδα της Ιαπωνίας και της Κίνας. Επίσης, οι Υπουργοί Εξωτερικών της, ε, της ΑΣΕΜ στο Δελχή συναντήθηκαν, ούτω ώστε να προετοιμάσουμε την ε, Σύνοδο Κορυφής που θα διοργανώσει η Ιταλία τον Οκτώβριο του 2014. Η σύνοδο κορυφή της Ιαπωνία. να σα πω λίγο το πλαίσιο, κανονικά είχε προγραμματιστεί το Μάρτιο του 2013, αλλά δυστυχώ η κυπριακή κρίση ξέσπασε τότε και έπρεπε να ακυρωθεί η σύνοδο κορυφή. Τότε κανονικά θα ξεκινούσαν διαπραγματεύσει για μια συμφωνία πλαίσιο που την ονομάζουν η Ιαπωνέζη Στρατηγική Εταιρική Συμφωνία, καθώς και για την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορίου, που ονομάζουν οι Ιαπωνέζοι Οικονομική ε, Συμφωνία Εταιρική σχέση. Αυτές οι διαπραγματεύσεις παρόλα αυτά ξεκίνησαν μετά τις 25 Μαρτίου, αλλά ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαμε για τις δύο προεδρίες να ξεκινήσουν και να συναντηθούμε τον ε, πρόεδρο Άμπε και να δούνε τι γίνεται μετά τις εκλογές ε, στη Γερουσία τον Ιούλιο, στην Ιαπωνία. Η Σύνοδος Κορυφής κράτησε μία ώρα και συνεχεία ακολούθησε το δείπνο. Ήταν μία ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό Άμπε να ε, ζητήσει στήριξη για τις βασικές πρωτοβουλίες για την αναζωγόνηση της ε, Ιαπωνέζικης οικονομίας, την ενίσχυση της ε, ασφάλειας, την πολιτική ορμή στις διαπραγματεύσεις για μια εταιρική συμφωνία στρατηγικής σημασίας, για κάποιες τομεακές συνεργασίες και για ανταλλαγή απόψεων για διάφορα θέματα ασφάλειας που συμπεριλαμβάνουν και βέβαια τα εδαφικά ζητήματα στην νοτιοανατολική Ασία. Επίσης ζήτησαμε από την Ιαπωνία να παίξει ηγετικό ρόλο για να συνεχίσει η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Μετά τη συνάντηση που έγινε στη Βαρσοβία των COP, όπου μειώθηκαν οι στόχοι, κατέβηκε η μπάρα. Ο... Παρουσιάστηκαν οι τρεις βασικοί άξονες της πολιτικής. Καταρχάς, ε, ε, το δημοσιονομικό, τα δημοσιονομικά κίνητρα, η ανάκαμψη της ε, οικονομίας και η εφαρμογή του τρίτου βέλουτς, όπως λέγεται, ε, οι οικονομικές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς εξηγήσαμε τις βασικέ μας πολιτικές για να εξασφαλίσουμε την μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και χαιρόμαστε για την θετική πολιτική του, του ΆΜΠΕ που αυξάνει την πιστοσύνη των καταναλωτών αλλά Θέλουμε να υπάρξουν διαρθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, που θα πρέπει να εφαρμοστούν νωρί σε αυτή την θητεία της ε, κυβέρνησης που θα έχει σχετική σταθερότητα. Ο πρώτος Μπαρόζο είπε ότι είχε συνόδους κορυφής τα τελευταία χρόνια με 7 διαφορετικούς ιαπωνέζου πρωθυπουργού. κάτι που δεν διευκολύνει βέβαια συζήτηση μεταξύ μα. Για την ασφάλεια, ο Άμπε ε, παρουσίασε το όραμά του για την Ιαπωνία. Ε, βασίζεται στην αρχή της διεθνούς συνεργασίας. Η Ιαπωνία θέλει να δημιουργηθεί ένα νέο ε, ε, Συμβούλιο Ασφάλειας, μια, να, κάποιες αναθεωρημένες γραμμές για την άμυνα και συνταγματική επανερμηνία, ούτως ώστε η Ιαπωνία να μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας. Επίσης, η Ιαπωνία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ε, στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ιαπωνία προ αυτήν την κατεύθυνση. Η Ιαπωνία βεβαίω θα πρέπει να λάβει υπόψη τι ευαισθησίε των γειτόνων τη που τις είδαμε κάτι στην τη της Κορέας. Το Τόκιο πρέπει να εξηγήσει πολύ σαφώς τι κάνει και ποιοι είναι οι λόγοι και τα κίνητρά του, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες από τους γείτονες της Ιαπωνίας. Επίσης, εμεί είπαμε ότι ενδιαφερόμαστε στην ασφάλεια της περιοχής και είπαμε ότι στη Σύνοδο ε, της Νοτιοανατολικής Ασίας θα θέλουμε να συμμετάσχουμε. Επίσης, ε, θέματα πολιτικής διαστήματος και κυβερνοασφάλειας μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Επίσης, πολιτική ορμή στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελευθερού εμπορίου και για την ε, συμφωνία πλαίσιο εταιρική σχέσης ε, για να πετύχει συμφωνία ελευθερού εμπορίου θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και στον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2013 ε, που μπήκε στην... Μια, είναι μια ρήτρα δηλαδή που μπήκε στην εντολή ε, είπαμε ότι δεν θα είναι θέμα ρουτίνας να αναθεώρηση ότι θα γίνει τον Απρίλιο και μιλήσαμε για τη σημασία ε, των οδικών χαρτών, ειδικά για τις ε, τους μη δασμολογικούς ε, φραγμούς, αλλά και για τις δημόσιες προμήθειες που συμφωνήσαμε με την Ιαπωνία όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Ο Πρωθυπουργό Άμπε είπε ότι η Ιαπωνία θέλει να ολοκληρώσει και τις δύο συμφωνίες μέχρι το τέλος του 2014 και ότι είναι αντίθετο στην σύνδεση που προτάθηκε μεταξύ της πολιτικής συμφωνίας και της εμπορικής συμφωνίας καθώς και στην πολιτική ρήτρα στην συμφωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, εξετάζουμε συνέχεια και στη διαπραγματεύση στον Καναδά, με την Αυστραλία και με την Νέα Ζηλανδία αυτό των ρητρών. Καθώ και με την Ιαπωνία βεβαίω. Όλοι ισχυρίζονται ότι δεν του αρέσουν αυτή η προσέγγιση από πλευρά μα. Είπαν ότι αυτή η προσέγγιση δεν ε, αρμόζει τις σχέσεις μας που βασίζεται, βασίζεται σε κοινέ αξίες και στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα και είπαν ότι πρέπει να αλλάξουμε τη θέση μας. Εξήγησαν την... Εμείς εξηγήσαμε τη θέση μας που είπα, και είπαμε ότι θα πρέπει βασικά, αφού έχουμε τις ίδιες ιδέες, να υποστρίζουμε στον άλλον, ούτω ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε πίεση σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται πολιτική πίεση. Αλλά δεν νομίζω ότι τους πείσαμε δεν πείσαμε τον Πρωθυπουργό Άμπε με, την, τα επιχειρηματά μας. Επίσης, ε, η συνεργασία για την ενέργεια, διαχείριση των κρίσεων, πυρηνική ασφάλεια και πυρηνική ενέργεια. Και είπαμε ότι η εταιρική σχέση έρευνας, ειδικά στα πλαίσια του ορίζοντα 2020, θα περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο. Το δείπνο, στο δείπνο συζητήσαμε διάφορα θέματα σοβαρά, δηλαδή ε, αστεία, Κίνα, η θάλασσα της Νότιας Κίνας, Βόρεια Κορέα, Μιανμάρ και Ρωσία, καθώς και η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Ο Πρωθυπουργό μίλησε για τις ανησυχίες της Ιαπωνίας, για τις εντάσεις που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία, όπου είπε ότι η Ιαπωνία έχει μια περιορισμένη αλλά σταθερή σχέση οι δράσεις της Κίνας στη θάλασσα και η προσπάθεια να αλλάξει το status quo θεωρούνται από τους Ιαπωνέζους ε, απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και επίσης είπε ότι αναγνωρίζει βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκοπεύει να άρει το εμπάργκο όπλων, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των εξαγωγών. Ε, οι Ιαπωνέζοι θέλουν να επανεκκινήσουν το διάλογο με την Κίνα και δεσμεύτηκαν να συζητήσουν με τους Κινέζους ηγέτες εν συνεχεία για αυτό το θέμα. Οι Ιαπωνέζοι είπαν ότι είχαν επαφές με το Ιράν. Σε αυτή τη φάση οι συζητήσεις ε, στη Γενέβη συνεχιζόταν ε, και οδήγησαν στο επιτυχές αποτέλεσμα που ξέρουμε. Οι Ιαπωνέζοι μίλησαν για τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργό τους όταν επισκέφθηκε τη χώρα και υποστήριξαν τις συζητήσεις α συν 3 για την αλλαγή του κλίματος. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που έχει η Ιαπωνία. Μετά τον μεγάλο σεισμό το 2011 και το κλείσιμο των πυρηνικών εγκαταστάσεων, είπαν ότι είναι υπέρ ε, ενός φιλόδοξου αποτελέσματος της διεθνής διαπραγματεύσεις και ότι θα πρέπει να έχουμε την πιο φιλόδοξη συμφωνία το 2015. Σε εκείνη τη φάση οι συζητήσεις στη Βαρσοβία συνεχιζόταν με τα αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε. Ε, στα πλαίσια των δύο συνόδων, της, συνόδου μάλλον κορυφής, ε, ε, ο πρόεδρος συναντήθηκε με τον ε, διοικητή της ε, Τράπεζας η Ιαπωνίας με επιχειρηματίες επίσης. Ενημέρωσε τους επικεφαλείς της ε, αντιπροσωπείας μας για τα αποτελέσματα. Ο Ντεχούχτ είχε διάφορες ε, υπουργικές συναντήσεις, ε, ειδικά για τα θέματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Αυτά συνοπτικά, Πρόεδρε, είναι όλα όσα διαμήθησαν στο Τόκιο. Νομίζω ότι συνολικά ήταν χρήσιμη και σημαντική η Σύνοδος Κορυφής, δίνει νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις, έγιναν κάποιες συζητήσει για μια ε, νέα σύνοδο που θα πρέπει να γίνει σχετικά ε, σύντομα, στο πρώτο μισό του 2014 και φυσικά τον Απρίλιο θα γίνει η αναθεώρηση ε, των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου και θα δούμε τότε τι γίνεται για την πολιτική συμφωνία. Του χρόνου θα είναι μια σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ιαπωνία ούτως ή άλλως. Και αν συμφωνείτε, θα περάσω τώρα στην Κίνα. Στην Κίνα. Ήταν η 16η συνάντηση κορυφής ε, Ένωση Ιαπωνία και δέκατη επέτειος της ε, σφαιρικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Μία, η πρώτη ευκαιρία που είχαν οι δύο πρόεδροι να, συναντήσουν τη νέα κινέζικη ηγεσία, αν και είχαν αντιμετωπίσει τους νέους ηγέτες χωρισμένα και σε διαφορετικά πλαίσια. Ο Πινγκ μας υπενθύμησε ότι ήρθε στις Βρυξέλλες το 2010 είδε τον ε, πρόεδρο Φαντρόμπ που ήταν πρωθυπουργός του Βελγίου και τον πρόεδρο Μπαρόσο που ήταν και τότε πρόεδρος της Επιτροπής. Έγινε αμέσω μετά η συνάντηση αυτή, την τρίτη ολομέλεια του κόμματο που μόλις είχε λάβει μια σειρά από σημαντικέ αποφάσεις που ακόμη προσπαθούμε να αναλύσουμε την πλήρη σημασία τους για το μέλλον των μεταρρυθμίσεων στην Κίνα. Ήταν λοιπόν κρίσιμη ε, ευκαιρία για να έρθουμε σε επαφή με τη νέα ηγεσία για να καταλάβουμε πού πάει η Κίνα. Προηγήθηκε την προηγουμένη μια συνάντηση και για πρώτη φορά δείπνο ε, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο Xi Jinping. Συνήθως μας καλεί ο Πρωθυπουργό, αλλά αυτή τη φορά είχαμε πολύ σημαντική συνεδρίαση που ξεπέρασε το χρόνο που προβλεπόταν και το δείπνο επίσης ξεπέρασε το χρόνο που είχε προβλεφθεί. Το πιο εντυπωσιακό ως μήνυμα είναι ότι η στάση τους ήταν πολύ θετική και επικοδομητική αλλά και πολύ διαφορετικό στυλ από τους δύο ηγέτες και δεν είμαστε οι μόνοι που το διαπιστώσαμε. Πολύ πιο άνετοι, πιο, πιο αυθόρμητοι, λιγότερη, λιγότερο διάβασμα από προετοιμασμένα κείμενα. Συνήθως τις προηγούμενες συναντήσεις κορυφής ήταν ε, ε, τις προηγούμενες φορές ε, στις συναντήσεις γενικά στην Ασία πολλές φορές έχεις την αίσθηση ότι δρούν με βάση σενάριο, ενώ τώρα υπήρχε περισσότερος αυθορμητισμός, αμεσότητα. Αυτοπεποίθηση βεβαίως από πλευράς τους, αλλά ήταν πολύ ανοιχτή για τα διάφορα θέματα που ήθελα να θίξουμε. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε θετικό κλίμα για την επόμενη φάση των σχέσεών μας, αυτή την πρώτη επίσημη επαφή σε ανώτατο επίπεδο. Υιοθετήσαμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό 2020 συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. συμφωνήσαμε σε αιτήσιο μηχανισμό αναθεώρηση. Δεν θα σα κρύψω οι διαπραγματεύσει ήταν σκληρέ για το θέμα αυτό. Τότε η αμεσότητα και η γενική αντιμετώπιση των ηγετών ε, δεν ήταν ε, ε, ίδιες με τη συμπεριφορά των ε, γραφειοκρατών. Κάναμε μάχες εκ του συστάνου για ένα κόμμα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι καλό. Είναι μια πιο θετική στρατηγική σχέση για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα συμφωνήσαμε την έναρξη διαπραγματεύσεων για διμερή συμφωνία επενδύσεων και επίσης να συζητήσουμε την αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων εμπορικών εντάσεων. Επίσης θα αναπτύξουμε νέους τομείς συνεργασίας, βιώσιμη ανάπτυξη και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία για ανταλλαγές ε, ατόμων. Όμως ε, έχουμε δυσχέρειες ε, για να προωθήσουμε την επίλυση των θεμάτων μετανάστευσης και προξενικών θεωρήσεων γιατί το αποτέλεσμα των συναντήσεων που είχαμε τον Οκτώβριο για το θέμα αυτό ήταν κάπως απογοητευτικό δεν ε, ήταν δυνατόν να αποφασίσουμε μια σύνδεση μεταξύ εξαίρεσης ε, προξενικών θεωρήσεων για διπλωμάτες και υποχρέωσης ε, επανεισδοχής. Θα συνεχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Οι δύο πρόεδροι εξέφρασαν ανησυχίε για εξελίξει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Ο Φαν Σημείωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο από πλευρά τη Κίνα, ιδιαίτερα στον τομέα των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά είπε ότι η πιστεύει ότι μπορεί να γίνει περισσότερο για να υπάρξει ελεύθερη έκφραση, ελευθερία του συνεταιρίζεστε και μειωνοτικά δικαιώματα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις, ε, το διάλογο για, για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συζήτησης για να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τις διαδικασίες για το θέμα αυτό. Ήταν πολύ επιτυχημένη η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου Λαμπρινίδη της Ένωσης για Ανθρώπινα Δικαιώματα το Σεπτέμβριο και προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερη όθηση και δυναμισμό σε αυτόν τον διάλογο που ορισμένε φορές είναι κάπως ε, τυπικές ανταλλαγές. Δεν θέλω να το κρύψω αυτό, αλλά θέλουμε να δώσουμε περισσότερη ενέργεια σε αυτές τις συζητήσεις. Οι συζητήσεις επίσης κάλυψαν εσωτερικές εξελίξεις, οικονομικά θέματα, εμπορικά θέματα, επενδυτικά θέματα και σχέσεων και διάφορα ε, συνολικά διεθνή θέματα. Αναπόφευκτα Ιράν, γιατί γίνονται συζητήσεις, Συρία, ε, θάλασσα της ε, Νότιας Κίνας και η Βόρεια Κορέα. Και για τα θέματα των διαμαχών τους με την Ιαπωνία για θέματα χωρικών υδάτων ε, μας είπαν είναι διμερεί θέματα να τα επιλύσουν οι χώρες ε, τις οποίες αφορούν. Όπως βλέπετε λοιπόν ήταν κάπως διαφορετικά τα μηνύματα που πήραμε από το Μπεϊτζίν και από το Τόκιο το θέμα αυτό. Η μόνιμη θέση μας είναι ότι και εμάς μας ενδιαφέρει και εμάς μας ενδιαφέρει η ευημερία και η ασφάλεια της περιοχής και εμάς μας ενδιαφέρει η ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά δεν παίρνουμε θέση για τις ε, αξιώσεις χωρικών υδάτων και τις εδαφικές αξιώσεις και καλούμε τις δύο πλευρές να διαχειριστούν την κρίση με κάθε μέσο και να προσπαθήσουν να βρουν λύση ιδιαίτερα στα πλαίσια των συζητήσεων μεταξύ της Κίνας και του ΑΣΕΑΝ για ένα δεχόμενο κώδικα δεοντολογίας. Όπως είπα, οι συζητήσεις για, την, για το θεματολόγιο 2020 ήταν κάπως δύσκολες και ολοκληρώθηκαν οι συζητήσει μόνο όταν ανακοινώθηκε και το αποτέλεσμα. Μετά αλλάξαμε βέβαια κάποια κόμματα και κάποιες ε, φράσεις και τελικά καταλήξαμε στη συμφωνία. Αλλά νομίζω, όπως είπα, ότι συνολικά είναι ισορροπημένο το αποτέλεσμα, αλλά είναι ζωντανό το έγγραφο αυτό. Θα το επικαιροποιούμε, θα το βελτιώνουμε στις ε, αλλεπάλληλες συναντήσεις κορυφής. Υπάρχει μια αναφορά στην ενδεχόμενη συμμετοχή της Ένωσης στις συναντήσεις Ανατολικής Ασίας. Αυτό ήταν ε, σημαντική πρόοδος, αν και η Κίνα επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση όλων για την ασφάλεια και την άμυνα. Σταδιακά θα ανεβάσουμε το επίπεδο του διαλόγου, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία για τη θαλάσσια ασφάλεια, ιδιαίτερα στον τομέα της αντιμετώπισης της πειρατείας. Εξετάζουμε τη δυνατότητα κοινών ε, ναυτικών γυμνασίων στον κόλπο του Άντεν του χρόνου. Αυτά είναι τα κυριότητα. Δεν θέλαμε να ξεκινήσει διάλογος για το κράτος δικαίου. Δεν καταφέραμε να αναφερθεί εκπεφρασμένα, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι είναι στοιχείο των πορισμάτων της Τρίτης Ολομέλειας. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο κείμενο. Αλλά υπάρχει μια αναφορά στην, στο θεματολόγιο 2020 σε νομικά και διοικητικά θέματα που νομίζουμε ότι ανοίγει την πόρτα για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Ιδιαίτερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Τέλος, για τις ανταλλαγές ατόμων συμπεριλαμβανομένες και της συνεργασίας, ε, για τις προξενήσεις, τους νέους, τη μετανάστευση, τον βιώσιμο τουρισμό και την, ε, τον πολιτισμό. Επίσης, εκφράστηκε δέσμευση να υπάρξει συνολική συμφωνία, γιατί οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται για γεωγραφικές ενδείξει. Να υπάρχει πρωτοβουλία συνεργασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να έχουμε διάλογο για την καινοτομία και τη συνεργασία και πολύ επιτυχημένη ε, ένα πολύ επιτυχημένο φόρουμ συνεργασίας για τα αστικά κέντρα όπου συμμετείχαν πολλοί ε, δήμαρχοι από τις δύο πλευρές και επίσης ε, ξεκινήσαμε έναν ετήσιο αναπτυξιακό διάλογο. Μια σειρά συμφωνίε υπογράφησαν. Μια διοικητική συμφωνία για συνεργασία στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, κοινή διακήρυξη για την ενεργειακή ασφάλεια και ένα γράμμα πρόθεση για την έρευνα και την καινοτομία συνεργασία στο επιστημιστικό τομέα, το γεωργικό τομέα και την βιοτεχνολογία. Ήταν πολύ έντονε συναντήσει. Είχαμε και αυτό το φόρουμ ε, για του επιχειρηματίε, για τι πόλει Καλύψαμε λοιπόν μια σειρά από θέματα. Νομίζω λοιπόν τη δέκατη επέτειος της ε, στρατικής μας σχέσης ε, ε, αποτέλεσε βάση για να φτιάξουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα για τις εξελίξεις στην επόμενη περίοδο. Υπάρχουν θέματα όπου έχουμε διαφορετικές απόψεις εμπόρια ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πρέπει να πω ότι συνολικά το κλίμα ήταν επικοδομητικό, θετικό. Οι διαφορές αυτές μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των ε, κοινών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλαγέ ε, στη δημογραφία και την τεράστια αστιφιλία που έχει να αντιμετωπίσει η Κίνα την προσεχή περίοδο, όπου η δική μας ε, τεχνογνωσία μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτά, ευχαριστώ, αλλά φυσικά στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες ή να ακούσω σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σάλιβαν για αυτή την ενδιαφέρουσα ενημέρωση που μας κάνατε. Θα ήθελα εάν να μάθω εάν οι, οι υπηρεσίες σας έχουν μια εκτίμηση του πώς πήγε ο πρώτος χρόνος ε, της νέας ηγεσία του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, ιδιαίτερα για το κοινωνικό θέμα, το ένα παιδί και των ε, στρατοπέδων επανα, επανεκπαίδευσης. Και κυρίως το κύριο στοιχείο αυτής της νέας πολιτικής ε, που είναι το οικονομικό, όπου αναφέρονται σε αποκέντρωση, ε, μάλιστα μιλάνε και για αποϋπουργοποίηση, δηλαδή ότι πολλές αποφάσεις δεν θα παίρνονται σε κεντρικό επίπεδο στα πλαίσια αυτά. Θα ήθελα να μου πείτε, εάν έχετε εκτίμηση, για το ότι οι νέοι ηγέτες της Κίνας έχουν καθορίσει ως στόχο είναι το 2020 να έχουν διπλασιάσει σε σχέση με το 2010 το ΑΕΠ και το μέσο εισόδημα. Κάτι άλλο. Το αναφέρατε στην εισαγωγή σας γενικότερο που αφορά τις σχέσεις με τον Καναδά. Στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα, παρουσιάσουμε την έκθεση, θα παρουσιάσουμε την έκθεση της συναδέλφου Ντέγκελ και συζητάμε αυτή τη στιγμή με ορισμένου συναδέλφου όπω τον κύριο Πέτερλε την έκθεση για την Κίνα. Και επίσης σήμερα έχουμε και την παρουσία κάποιων ε, νομοθετών από τις ΗΠΑ. Κύριε Σάλιβαν, ο Σάλιβαν, θέσατε τα θέματα που, θέτει, που θέτουν οι συμφωνίες αυτές σε σχέση με την δημοκρατική ρήτρα. Πώς ως Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, πώς ως Επιτροπή θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα γιατί πρέπει να κάνουμε το παιδαγωγικό μας καθήκον, να ε, καταδείξουμε στους εταίρους μας ότι η δημοκρατική ρήτρα έχει αμοιβαίο χαρακτήρα. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να απαιτηθεί και από τους δύο. Πώς λοιπόν θα παρουσιάσετε το θέμα αυτό, με ποιο κέντρο βάρους, γιατί από ό,τι φαίνεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ ε, έχει υπάρξει μια δημιουργική λύση λέγοντας ότι θα βάλουμε ε, στα απορίσματα της συμφωνίας ότι εμπλεόμεθα από κοινέ αρχές και θα τις ακολουθήσουμε. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι θα κάνουμε σαν συμφωνίες για το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι του ανησυχεί και θα ήθελα να μάθω τι θα γίνει. Διότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι σε καμία περίπτωση μια τέτοια ρήτρα δεν θα έπρεπε να τους δημιουργεί ανησυχίε, γιατί είναι χώρες που έχουν ε, υψηλό επίπεδο δημοκρατικής ε, ανάπτυξης. Ο κύριος Τάνοκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που είσαι εδώ, David, μαζί μα, ε, Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι στρατηγικές συναντήσεις και ανακύπτουν διάφορες ερωτήσεις. Καταρχάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, η ιδέα μια ζώνη μιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου, πώς ταιριάζει αυτό στην μακροπρόθεσμη στρατηγική της ε, ε, στρατηγικής με την άλλη πλευρά του ειρηνικού και κυρίως σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο πλαίσιμο, μια συμφωνία ελευθερίου εμπορίου που θα φτάσει από τη Βόρεια Αμερική μέχρι τη Λατινική Αμερική, το Μεξικό, Καναδά, ΗΠΑ και μετά θα περάσει στον ελληνικό στις μεγάλες δημοκρατίες ε, όπως η Ιαπωνία. Ε, έτσι σκέφτεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ε, διάστημα. Κατά δεύτερον, τι πιστεύετε για την οικονομία της Ιαπωνίας, λειτουργεί η οικονομία τους, ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, ό,τι αφορά την ε, λειτουργικότητά της και πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας πριν από κάποιες χρόνια. Υπήρχε αυτή η ιδέα της προσέγγισης, της προσέγγισης. Τώρα φαίνεται ότι έχουν ψυχρανθεί και πάλι σχέσεις. Έγιναν πριν από κάποιες ε, ημέρες, ημέρες κάποιες δηλώσεις ανησυχητικές από πλευρά της Κίνας σε ό,τι αφορά τις περιοχές αυτές που είναι υποκλητικές οι δηλώσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιδράσει ή κάθε άστον έχει προβεί σε κάποια δήλωση γιατί αυτό ενδεχομένως να είναι ένα σημείο καμπής και αν ε, ξεσπάσουν εχθροπραξίες μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων, αυτό θα έχει ευρύτατε συνέπειες όχι μόνο για την περιοχή της ε, Απανατολής, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να πω ότι είμαι πρόεδρος της Επιτροπής ε, για τις σχέσεις με την Ταϊβάν που και αυτή είναι ε, εμπλεκόμενος φορέας και οι άλλοι δύο χώρες ασφαλώς. Αλλά η PRC εκεί να φαίνεται ότι έχει αξιώσει σε ό,τι αφορά χωρικά ύδατα, έχουν λάβει αποζημιώσει ε, από την ε, Φιλιππίνη και με το Βιετνάμ είναι πολύ αυστηρέ ε, και στο Βιετνάμ έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση και αναφερθήκατε και στον ΑΣΕΑΝ. Θα ήθελα να μα διευκρινίσετε τον ρόλο του ΑΣΕΑΝ. Πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί ένα κώδικα θεαντολογία επίση, σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν και τον πρόεδρο εκεί δεν φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει μια μεγάλη κίνηση προ την κατεύθυνση αυτή. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω στο πιο εγχώριο μέτωπο. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα πρόκειται να εναρμονίσει τις ε, θεωρήσεις για την ε, Κίνα. Ε, αν στην Κίνα παίρνει κάποιος βίζα Σέγγεν να μπορεί να εισέλθει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα γίνει διμερός από το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά και τις διαπραγματεύσεις ε, με την πρεσβεία, γιατί χάνει στην παρούσα φάση μερίδεο από την κινέζικο τουρισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το λύσουμε ως πρόβλημα. Ιδάλλως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει διαφορετικό σύστημα Σέγγεν και το χρειαζόμαστε ασφαλώς αυτό γιατί είναι σημαντική αυτή η εταίρη. Προφανώς όμως αν έχει κάποιος βίζα Σέγγεν θα πρέπει να μπορεί σχετικά εύκολα να επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρόεδρος δεν μιλάει. Σχολιάζει ο κύριος Άτκινς η καρέκλα του Πρόεδρου. Σας ευχαριστώ κύριε Σέλβαν που ήλθατε να μας μιλήσετε, να σχολιάσω και τις δύο σας ε, παρουσιάσεις μετά από αυτά που είπε και ο Τσάλς. Πείτε μας δύο-τρία στοιχεία για το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία. Καταρχάς, Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την Κορέα, τη Βόρεια Κορέα ιδιαίτερως και την Ιαπωνία και κατά δεύτερον έγιναν συζητήσεις καθόλου για το πρινικό ατύχημα στην Ιαπωνία και το τι επιπτώσεις είχε αυτό στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την Κίνα τώρα. Δύο πτυχές θα ήθελα να τονίσουμε και να τονίζουμε διαρκώς. Καταρχάς, την Ιαπωνίδη στη θέση της ε, Κίνας στο Ηνωμένο, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ε, Συρία. Εδώ θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πιο πολύ πίεση. Άραγε, εγώ θα έλεγα ότι δεδομένη τη κατάσταση ε, στη Συρία, μάλλον η κατάσταση στη Συρία προκαλείται και συνεχίζεται λόγω της Ρωσίας και της Κίνας ε, εν μέρη. Με δεύτερο σημείο που με ανησυχεί. Σημειώσαμε πως η Κίνα κινούνται μέσα στην Αφρική σε εμπορικά θέματα, πολύ δυναμικά και φαίνεται ότι υποστηρίζει διαρκώς κάποιες ε, από τις χειρότερες αφρικανικές δικτατορίες. Πολύ απλά επειδή έχει οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα. Αυτό είναι άραγε κάτι το οποίο θα έπρεπε τακτικά να το αναφέρουμε, να κάνουν εμπόριο με ποιον θέλουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν επιπτώσεις όταν ε, Μιλάμε για κάποιε συγκεκριμένε κυβερνήσει ανάλογα και με τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων και ίσω θα έπρεπε να τοποθετηθούμε κι εμεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. I give the floor to Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιαμόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που θα να κάνω ε, τέθησαν από τους προηγούμενους. Όπως βλέπετε, ε, λόγω των ε, σχέσεων που έχουμε με τις δύο χώρες, ε, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η ένταση με, λόγω των ελέγχων που κάνει η Κίνα σε ορισμένα νησιά. Επίσης και οι δύο συνομιλητές, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμφωνία που έχουμε με τις ΗΠΑ, TTIP. Και επίσης, πώς εκτιμούν οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναφτιάχνουμε στην ουσία την Οικονομική Ένωση για να είναι στο επίπεδο της Νομισματικής Ένωσης. Ε, τους ενδιαφέρουν αυτές οι αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. κύριο Σόλτς είναι ο τελευταίος ομιλητής στο κατάλογο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σάλιβαν για την ε, καλή του ενημέρωση. Τρεις ερωτήσεις σύντομες. Μιλήσατε για τη συνεργασία για τα ενεργειακά κλάστερ. Έχει διαδραματίσει αυτό συγκεκριμένο ρόλο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις δύο πλευρές, τη συνεργασία σε ό,τι αφορά και την περιβαλλοντική κατάσταση στην Κίνα, γιατί προχωράμε και έρχεται ο χειμώνα, ξέρετε, και ασφαλώς είναι μεγάλη πρόκληση. Τι σημαίνει αυτό όμως συγκεκριμένα αυτή η συνεργασία για τα ενεργειακά κλάστερ, σε ό,τι αφορά επίσης την απόδοση των οικονομικών φορέων, σε ό,τι αφορά την Κίνα. Δεύτερη ερώτηση. Ο ρόλος της συνεργασία ε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, ε, της ε, συνάντησης στα πλαίσια του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά και τις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις. Έχετε πιο πολλές λεπτομέρειες και υπήρξε πιο εις βάθος συνεργασία σε ό,τι αφορά την σύνοδο. Ύστερα το θέμα του NSA. σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη Σύνοδο στις συνομιλίες που έγιναν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη γερμανική πρωτοβουλία στα πλαίσια του ΟΗΕ για ένα ψήφισμα για την ιδιωτική σφαίρα από πλευρά του ΟΗΕ και κατά πόσον αυτό θα ίσχυε και για άλλες χώρες, κατά πόσον προσυπογράφεται αυτή την προσέγγιση. σα ευχαριστώ. Τελευταία ο Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ε, συγχαίρω και για την πραγωγή σας. Ε, κύριο Σάλιβαν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, καλή σας παρουσίαση. Μία σύντομη ερώτηση να σας κάνω. Από ό,τι φαίνεται η κινέζικη πλευρά ανησυχεί. Αναρωτιέται τι σημαίνει και ποιε θα είναι οι συνέπειε του TTIP. Το θέμα αυτό τη Ιταλική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων. Αυτό τέθηκε στη Σύνοδο ω θέμα. Και πώ εκτιμάτε τι ανησυχίε αυτέ από πλευρά τη Κίνα και κατά πόσο μπορούμε να απαντήσουμε και να καθισχάσουμε τι ανησυχίε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. δεν ήθελε κανεί άλλο να πάρει το λόγο. Να δώσω λοιπόν το λόγο και πάλι στον κύριο Σάλμα να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές για τις αριθμές ε, και λεπτομέρειες ε, ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Μιλαμόν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ξεκινήσω από αυτό. Και ο πρόεδρος ε, Φαρόμπουη και ο πρόεδρος Μπαρόζο και στις δύο συνόδους κορυφής μίλησαν διαμακρών για την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Παρουσίασαν έναν υφάλιο μήνυμα κάποιων μετριοπαθών βελτιώσεων, σταθεροποίηση κατάστασης και κάποιων προοπτικών για βελτίωση, χωρίς να προσπαθήσουμε να ε, υπερβάλλουμε, ας πούμε, ούτε τις προκλήσεις, αλλά ούτε και τις βελτιώσεις. Και οι δύο πρόεδροι μου είπαν ότι αυτό που είναι εντυπωσιακό και στις δύο συνόδους κορυφής είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ανησυχίας για την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη που παρατηρούσαμε πριν από ένα χρόνο ή πριν δύο χρόνια. Υπάρχει έτσι μια εντύπωση ότι η διεθνής κοινότητα έχει δεχτεί ότι η Ευρώπη έκανε διάφορα πράγματα για να βελτιώσει την κατάσταση, να αντιμετωπίσει την κρίση και ότι είμαστε σωστή πορεία. Ας μην είμαστε αυτάρες και υπάρχουν πολλές προκλήσεις ακόμα και ούτε θα εφησυχάσουμε βέβαια. Αλλά δεν δίνεται πια τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη για διαβεβαιώσει από πλευρά μα, για την οικονομική μας κατάσταση. Γενικά υπάρχει μια αποδοχή ότι η Ευρώπη έκανε πολλά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια, έκανε τα δύσκολα πράγματα που έπρεπε να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η κρίση και τώρα είναι σε πολύ καλύτερη πορεία. Για το θέμα του κύριου Σαλαφράγκα, για την Ολομέλεια και τις μεταρρυθμίσεις. Ακόμα μελετούμε το θέμα αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ας μην συνάγουμε βιαστικά συμπεράσματα μόνο μετά από ένα έγγραφο. Γιατί σε αυτές τις χώρες τίποτα δεν είναι όπως αυτό που λένε τα έγγραφα. Ένα πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι το μήνυμα στην Κίνα, το μήνυμα που έδωσαν οι ηγέτες, είναι ότι πρόκειται για μια νέα ουσιαστική βαθιά μεταρρύθμιση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική του ενός παιδιού, την κατάργηση της, των στρατόπεδων επανεκπαίδευσης, ε, μια μεγαλύτερη απελευθέρωση της, του δικαιώματος μετακίνησης στη χώρα. Ο πρόεδρος ε, μίλησε για τις προκλήσεις που υπάρχουν ε, των μετακινήσεων από την ύπεθρο της πόλης, αυτή η αστιφιλία ε, δεν θέλει η Κίνα να δημιουργήσει τεχνικέδου πόλεις ε, στις πόλεις, ε, όπως έχουμε δει στη Λατινική Αμερική Φερρυπίν. Δεν θέλει με την πολιτική της να δώσει κίνητρα σε μια τέτοια κατάσταση. Επομένως υπάρχει αίσθηση ότι κάτι γίνεται για αυτά τα θέματα στην Κίνα. Υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα. Επίσης, ε, στο οικονομικό επίπεδο ε, είναι πολύ μεγάλο θέμα η μεταρρύθμιση των, οικονομικών, των ε, κρατικών επιχειρήσεων, που ήταν μεγάλο άχθος. Όλα αυτά τα χωνεύουμε λοιπόν και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Με την εφαρμογή δηλαδή. Πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Αυτά που μας είπαν οι ηγέτες όμως της Κίνας είναι ότι είναι ένα σημαντικό πακέτο μεταρρυθμίσεων που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αυτό το θέμα της μετακίνησης από την ύπεθρο της πόλης, ε, μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ε, η πρόκληση Ανατολής και Δύσης, δηλαδή η υπερβολική ανάπτυξη της Ανατολικής Κίνας και η ε, καθυστέρηση που υπάρχει στη Δυτική Κίνα, υπάρχει πραγματικά ένα πλήρες πακέτο μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές πολιτικές μεταρρυθμίσεις, εκεί όλοι συμφωνούμε. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι προς το παρόν υπάρχει πρόθεση να γίνει μια ουσιαστική αλλαγή ε, στην πολιτική κατάσταση. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί βέβαια στο μέλλον. Με ρωτήσετε για το θέμα των ουσιαστικών ρητρών στις συμφωνίες μας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα και απλά. Ξέρετε ότι έχω μια ισχυρή εντολή να επιμείνουμε σε πολιτικές ρήτρες. Στι συμφωνίες μας και να επιμείνουμε στη σύνδεση, στη διασύνδεση ανάμεσα στι πολιτικές συμφωνίες και στις εμπορικές ή τομεακέ συμφωνίες. Και ξέρετε γιατί το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι τομεακέ συμφωνίες υπόκεινται πάντα σε, κάποιες, σε κάποιους πολιτικούς όρους και προποθέσει. Αν α πούμε, δεν εμπιστευόμαστε μια χώρα ότι μπορεί να σεβαστεί ας πούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τι πολιτικέ προποθέσει τότε θα έχουμε πάντα τη δυνατότητα να αναστείλουμε τι συμφωνίε. Αυτό είναι σαφέ. και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Για πολλού εταίρου μα, η ιδέα ότι εμεί του επιβάλλουμε τέτοιε ρήτρες, ότι του ζητάμε να δεχτούν αυτέ τι ρήτρες, θεωρείται προσβλητική. Προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε ότι αυτό είναι αμοιβαίο, ότι και εμεί θα δεχόμαστε κάτι τέτοιο, θα δεχόμαστε την ίδια ευθύνη. Αλλά το θεωρούν εντελώ απαράδεκτο. Εμείς προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι για μας είναι ε, υπάρχει η εξής πρόκληση. Ότι αν κάνουμε εξαιρέσει, πού θα σταματήσουμε στο μέλλον. Γιατί θα γίνει μια συζήτηση για με κάποιες χώρες, ποιες θα δεχτούν αυτές τις ρήτρε, ποιες θα πρέπει να εξαιρέσουμε, ποιες όχι κτλ. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε βρει τρόπο να πείσουμε τους εταίρους μας ότι αυτή είναι μια καλή ιδέα, ιδέα των ρητρών. Προσπαθούμε τώρα να διερευνήσουμε λιγάκι τα επιχειρήματα, τη φρασιολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε μήπως μπορούμε να υπερκεράσουμε το πρόβλημα. Ειδικά με τον Καναδά, ας πούμε, ε, που υπάρχει περίπτωση, να είναι η πρώτη περίπτωση επιτυχούς εμπορικής ε, διαπραγμάτευσης ε, ή διαπραγμάτευσης πολιτικής συμφωνίας. και το Συμβούλιο που αποφάσισε ομόφωνα αυτή τη θέση θα πρέπει να καταγράψει το θέμα αυτό. Αλλά δεν έχουμε παραδοθεί ακόμα, δεν έχουμε πελπιστεί ότι μπορούμε να βρούμε κάποια επιχειρήματα που μπορεί να πείσουν α, τους εταίρους μας που έχουν τις ίδιες απόψεις και αξίες ότι μπορούμε τέλος πάντων να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Αλλά πάντως είναι δύσκολο το θέμα. Για τα άλλα ερωτήματα που ακούστηκαν, ειδικά για το εμπόριο και στις δύο περιπτώσεις και για την Ιαπωνία και για την Κίνα η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων ε, δεν αναφέρθηκε ρητά, μόνο εν παρόδο. Δεν θεωρείται πρόβλημα. Η Ιαπωνία τονίζει ότι η δέσμευσή της στην, ε, στις διαπραγματεύσεις δεν μειώνει τη δέσμευσή της για ε, συμφωνία ελευθερου εμπορίου μαζί μας. Κύριε Τάνοκ, για αυτό που με ρωτήσατε εσείς, Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ελπίζουμε, και ο κ. Σόλτσμαν το είπε για τον ΠΟΕ, μοιάζει ότι θα υπάρξει ε, ε, επιτυχής κατάληξη στη διάσκεψη του Μπαλί και θα υπάρξει κάποια ε, περιορισμένη πρόοδος στην ατζέντα της Ντόχα, που θα ήταν ευπρόσδεκτο. Ξέρετε ότι τα πολυμερή αποτελέσματα, οι πολυμερείς καταλήξεις είναι πολύ καλύτερες από τα, τις αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ο ΠΟΕ θα είναι σε θέση να φτάσει σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία για το εμπόριο. Επομένως θα συνεχίσουμε τις διμερείς ε, διευθετήσεις, αλλά συμφωνούμε κύριε Τάνοκ ότι αν οι, οι ασιατικές χώρες έχουν μια δική τους συμφωνία εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, αν εμείς έχουμε με το Μεξικό, με τη ΣΥΠΑ και με τον Καναδά, όλα αυτά αρχίζουν τελικά να κολλάνε και να δημιουργούν ένα μοσαϊκό όλες αυτές οι ψηφίδες. Μπορεί κάποια στιγμή λοιπόν όλοι να ξαναπάμε στη Γενέβη και όλα αυτά όλες αυτές τις ψηφίδες να τις βάλουμε σε ένα πλαίσιο πούμε και να φτιάξουμε ένα πολυμερές πλαίσιο. Εκεί όμως είμαστε ακόμα. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την περιοχή, είναι δύσκολες. Υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα εδαφικών διενέξεων, κάποια αίσθηση ιστορικών δικαιών Στην Ασία υπάρχει μια περιοχή, είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται οικονομικά. Υπάρχει μια αλληλεξάρτηση οικονομική των χωρών, αλλά υπάρχει μια ευάλωτη ασφάλεια, θα έλεγα. Η αίσθηση ασφάλειας. Και οι εντάσεις που δεν τις αντιμετωπίζουμε σωστά μπορούν να οδηγήσουν σε διενέξεις, σε συγκρούσεις, σε σειράξεις. Και το ξέρουμε αυτό από την εμπειρία μας στην Ευρώπη. Ε, ορισμένοι μιλάνε για μια νέα αρχιτεκτονική για την ασφάλεια στην Ασία, ούτω ώστε όλες αυτές οι διαφωνίες να διευθετηθούν διπλωματικά και όχι με διμερείς διενέξεις. Υπάρχουν πολλές εντάσεις. Οι σχέσεις μεταξύ ε, Ιαπωνίας και Κορέας δεν είναι πολύ καλές. Οι σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας είναι τεταμένες και υπάρχουν και εντάσεις μεταξύ Κίνας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ΑΖΕΑΝ είναι σημαντικός πυλώνας ε, και υποστηρίζει και την πολιτική μας στην περιοχή. Και ένας κώδικας διοντολογίας θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα για μια ευρύτερη αρχιτεκτονική για την ασφάλεια. Κύριε Τάνο, και το θέμα των θεωρήσεων. Δεν ξέρω στην πράξη πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Το καλύτερο θα ήταν, μα ε, να σας πω την προσωπική μου γνώμη βέβαια, να μπείτε εσείς και η Ιρλανδία α, στο Σέγγεν. Τότε θα χρειάζεται να κουβαλάω και το διαβατήριό μου κάθε φορά που θα πάω στην πατρίδα μου. Είναι η μοναδική περίπτωση που κουβαλάω το διαβατήριό μου. Καλό θα ήταν να είχαμε επίσης ένα κοινό καθεστώς θεωρήσεων και για τα 28 κρατημέλη. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτό, τουλάχιστον οι εθνικές θεωρήσεις και οι θεωρήσεις Schengen θα μπορούσαν να χρησιμεύουν η μία αντί της άλλης. Καλό θα ήταν αυτό. Και καλό θα ήταν και για τους εταίρους μας εξάλλου. Σε Ρόμπερτ, μίλησα για την Ιαπωνία και την Κορέα, για το πυρηνικό ατύχημα. Είναι σαφές ότι η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τεράστιο, τεράστιες προκλήσεις στην ενεργειακή πολιτική και αυτό απεικονίζεται δυστυχώς και στη μείωση των μεσοπρόθεσμων στόχων τους ε, για τις εκπομπές. Δεν έχουν σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν με ασφάλεια πολλές από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Τόνισα ότι και πέρασα ένα μήνυμα ότι θεωρούμε την Ιαπωνία σύμμαχό μας στις διαπραγματεύσεις ΚΟΠ του ΟΗΕ και δεν θα πρέπει η ε, κατάσταση που αντιμετωπίζουν ε, να υποσκάψει τη δυνατότητα για φιλόδοξα αποτελέσματα. Για τη Συρία. Στις, ε, στις συζητήσεις πάντα είχα την αίσθηση ότι όταν συζητάμε την Συρία με την Κίνα, βασικά συμφωνούμε, εκτός από το τελευταίο κομματάκι. Του τι κάνουμε τώρα. Συμφωνούν με όλε τι αναλύσει. Από το συμπέρασμα του ποιο είναι. Όχι. Δεν πρέπει οι, οι άλλοι να παρέμβουν. Δεν, πρέπει, δεν βοηθάει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλή κατάσταση. Λυπούμαστε. Από την άλλη θέλω να τονίσω ότι η Κίνα είναι πολύ επικοδομητικό εταίρος στις συζητήσεις ε, για το Ιράν. Η κάθε Άστον είπε δημόσια ότι η Κίνα ήταν πολύτιμος εταίρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν και έπαιξε πολύ θετικό ρόλο. Επομένως δεν είναι σωστό να λέμε ότι συνολικά ας πούμε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις ε, σχέσεις μας με την ε, Κίνα, αλλά η Συρία είναι τεράστιο σημείο διαφωνίας. Και βεβαίως οι ανθρωπιστικές συνέπειες του τι συμβαίνει στη Συρία είναι δραματικές για την Αφρική. Συμφωνήσαμε να έχουμε έναν αναπτυξιακό διάλογο και να συζητήσουμε όλα τα αναπτυξιακά θέματα. Έχετε δίκιο ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις μεταξύ ημών και εκείνων και εμείς θα πρέπει να βασιστούμε ε, στις δικές μας απόψεις, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Κάποιες αφρικανικές χώρες αρχίζουν να καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνουν ότι η εμπλοκή της Κίνας δεν είναι αμερικός τους και θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση στο μέλλον. Αλλά η Κίνα θα είναι σημαντικός εταίρος, σαφώς, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά στην Αφρική, και θα πρέπει να συνεργαστούμε όσο πιο επικοδομητικά μπορούμε με τους Κινέζους για την ενέργεια. Ξέρω ότι ίσως είμαι λίγο φλίαρος, αλλά θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω σιγά σιγά. Στο πακέτο 2020 που συμφωνήσαμε με τους ε, Κινέζους, υπάρχει και ο ενεργειακός διάλογος, όπου μιλάμε για την ε, παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, ε, εξετάζουμε και νομοθετήματα για την ενέργεια, πρότυπα, διατυπώσεις, συνεργασία για τεχνολογίες με χαμηλό άνθρακα, χαμηλές εκπομπές, διοξιδίου του άνθρακα και ενίσχυση των εργασιών για ένα ε, ευρωπαϊκό-κινέζικο κέντρο καθαρής ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης των θεμάτων της ανάπτυξης πυρηνικών εγκαταστάσεων με ασφαλή τρόπο σε μια συμφωνία Euratom με την Κίνα. Και το τελευταίο σημείο είναι η ενίσχυση της συνεργασίας για την ρύθμιση και νομοθεσία της ενέργειας ε, με εφαρμογή των των πρακτικών. Όλους αυτούς τους τομείς του συζητήσαμε. Αυτό που θα θέλαμε να συζητήσουμε στη Σύνοδο δεν το θέλησαν οι οι Κινέζοι είναι η πράσινη ανάπτυξη σε ένα ασφαλή κόσμο. Γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά κοινά σε αυτά τα θέματα τη ε, πράσινη ε, ανάπτυξη. Και ξέρετε πολύ καλά, σωστά είπατε, ότι όποιο έχει επισκεφτεί την Κίνα και ειδικά το Πεκίνο, ξέρουν, ξέρει πόσα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Και εξάλλου το αναγνωρίζει και ο κινέζικος πληθυσμός αυτό. Και καταλαβαίνει πια ότι πρέπει να ανταποκριθούν και να λάβουν υπόψη τους ε, τα προβλήματα και υπάρχει και στο πρόγραμμα της Τρίτης Ολομέλειας. Καμία αναφορά όμως δεν έγινε στα θέματα της ιδιωτικής σφαίρας και στην προστασία των δεδομένων. Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και αν παρέλειψα κάτι, εάν, ή αν θέλετε κάποια ειδική πληροφορία, μπορούμε να το δούμε και διμερώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Ο κύριος Βημόν δυστυχώς στις 12.30 μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει. Ε, ίσως υπάρχει κάτι το επίγον ε, σε σχέση με την συνάντηση κορυφής στο Βίλνιους. Τα πάντων, ατυχία. Αλλά και για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο Ντέβιντο Σάλιμαν, που είναι ο εκτελεστικό γενικό διευθυντή. Και ευχαριστώ και την παρουσία τη Προεδρία, τον κύριο Καρόμπλη. Ίσως λοιπόν και οι δύο θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε την ε, παρουσίασή σας. Ξέρουμε ότι μια σειρά από προτάσεις που έχει κάνει το Κοινοβούλιο Ε, ε, έχει απόψεις που τη σημερίζεται και η κυρία Άστον. Μας ανησυχεί ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις ε, σωστές στη σκέψη, στην έκθεση συγγνώμη, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Διότι αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να εκλεγεί το νέο κοινοβούλιο, η νέα επιτροπή και η νέα ύπατη ή ο νέος ύπατος εκπρόσωπος θα χάσουμε άλλα δύο χρόνια. Όμως έχουμε ήδη πιστεύω τη βάση για να προχωρήσουμε σε μια σειρά από θέματα. Να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλά στην, ε, στα 3,5 χρόνια της ε, ε, ανάπτυξης δραστηριότητας. Ε, μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το ποτήρι είναι το μισό γεμάτο. Αλλά ε, πρέπει να γίνουν πολλά και στο δεύτερο τμήμα της θητείας Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε περισσότερο με την εφαρμογή. Και ε, θα θέλαμε να είστε λίγο πιο φιλόδοξοι παρακαλώ για να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. Βλέπουμε ότι τα σημεία όπου διατυπώσαμε επικρίσεις, δηλαδή ότι πρέπει να βελτιωθεί η σχέση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στα σημεία αυτά και ότι επίσης ότι είπα ότι η εκπρόσωπος πρέπει να αναλαμβάνει περισσότερο το ρόλο της ως αντιπροέδρου της Επιτροπής για να μπορεί να παίζει και η Επιτροπή το ρόλο της και ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να δημιουργηθεί γύρω από την Αντιπρόεδρο η αναγκαία κρίσιμη μάζα για να μπορέσει να προχωρήσει. Είναι λοιπόν σημαντικό για να έχουμε και τις αναγκαίες ε, συνεργίες ούτω ώστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να έχουν αποτέλεσμα και αυτές οι συνέργειες. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα θέματα για το κέντρο αντιμετώπισης ε, των επιγουσών κρίσεων που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της συνθήκης, με το θέμα των ε, αναπληρωτών ούτως ώστε να αποφεληθούμε από τα λάθη που έχουν γίνει ε, για τη δεύτερη θητεία. και να προετοιμαστούμε για τη συνάντηση για θέματα άμυνα το Δεκέμβριο για να υπάρξει διαρθρωμένη συνεργασία. Και αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει τώρα. Είναι μόνο παραδείγματα. Θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι οι υπάλληλοι της Ένωσης είναι οι απλοί στρατιώτες και εκπρόσωποι των κρατών οι αξιωματικοί και στρατηγοί. Τα κράτη-μέλη νομίζουν ότι 30% της τελέχωσης πρέπει να προέρχεται από τα κράτη-μέλη και ότι αυτοί πρέπει να είναι πάντα οι υψηλόβαθμοί. Όχι, εμείς νομίζουμε ότι το 30% αυτό πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Αυτό μοιάζει να έχει παγιωθεί. Και αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι της Ένωσης δεν μπορούν να ε, προαχθούν. Και αυτό δημιουργεί απογοήτευση. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι μόνο παραδείγματα που θέλω να αναφέρω, παραδείγματα θεμάτων που μας ε, ανησυχούν. Νομίζω ότι έχουμε και τη διαπραγματεύση για τον προπολογισμό. Ο κύριος Σαλαφράγκα μπορεί να μας πει επίσης ε, τι θα γίνει με τον προπολογισμό των ειδικών αντιπροσώπων. Βλέπω δηλαδή γιατί όλοι αυτοί σχετίζονται με το Συμβούλιο, γιατί δεν είναι στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης η Επιτροπή ε, ούτε καν την ε, πολιτική γειτονία δεν μοιάζει να είναι σε θέση να κάνει. Όλα αυτά θέλουν να τα κάνει η εξωτερική δράση, τα κράτη-μέλη. Αλλά μετά διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένου τομεί ε, όπως των ειδικών αντιπροσώπων προτιμούν να είναι στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη. Από την άλλη μεριά όμως οι ειδικοί αντιπρόσωποι θεωρούνται και σαν πρέσβει των ε, κρατών μελών. Άρα υπάγονται από τη μία στο Συμβούλιο και από την άλλη στην Επιτροπή. Και αυτό έχει να κάνει και με την αύξηση του κόστους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από σημεία και ανέφερα μόνο ορισμένα ε, όπου μας εκπλήσει που δεν έχουν ε, συντελεστεί αναγκαίες αλλαγές. Και μπορώ να σα υποσχεθώ ότι και το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει την ίδια άποψη αν δεν γίνουν αυτέ οι διαρθρωτικέ αλλαγέ. Αν δεν γίνουν αυτέ οι διαρθρωτικέ αλλαγέ, μπορεί να υπάρξει και θέμα προπολογισμού. Γιατί όλα αυτά είναι κατά της, συνθήκη συνθήκης και κατά των συμπεμονηθέντων. Ήταν υποχρεωτική η στόχη αυτή. Θα σκεφτούμε τι πολιτικά μέσα θα αξιοποιήσουμε εάν αυτοί οι συμπεφωνημένοι στόχοι δεν γίνουν σεβαστοί. Δεν είναι δυνατόν ε, τα κράτη-μέλη να θεωρούν ότι η υπηρεσία εξωτερική δράση είναι απλώ άλλο ένα τμήμα των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών του. Αυτά είναι ισόδη θέματα για μας. Θέλουμε να είναι δυνατόν Ε, να μην είναι δυνατόν. Συγγνώμη, να είναι δυνατόν ένας ε, εθνικός ε, υπάλληλος να είναι στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, εάν είναι ικανοποιητική η απόδοσή του. Διότι αν δεν υπάρχει δυνατότητα θα υπάρχουν πάντα θέματα που ανήκει ο καθένας. Και αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιες για θέτουν το θέμα του πόσο πιστός είναι κάποιος σε μια υπηρεσία. Ξέρετε ότι υπάλληλοι είναι και αυτοί άτομα και φέρονται ως άνθρωποι. Οι αποφάσεις που να παίρνουμε ως Ένωση δεν επιτρέπονται. Αν θέλουμε λοιπόν κάποιος σε μέσο επίπεδο βαθμού αποφασίσει να έρθει στην Ένωση και μετά θέλει να μείνει να μπορεί να γίνεται. Αν είμαι νέος υπάλληλος από την άλλη μεριά και μετά πρέπει να ανακοινώσω στο κράτος μέλο μου, ενώ είμαι νέο υπάλληλο αυτό το κράτος μέλος, στο οποίο θα επανέλθω, κάτι το δυσάρεστο για αυτό που συνέβη. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να γίνει κάτι για αυτό το θέμα και ελπίζω οι αρμόδιοι της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης να έχει ε, περισσότερο θάρρος να κάνει αυτές τις αλλαγές. Γιατί αλλιώ ε, όσοι θα του διαδεχτούν θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουν αυτό. Ξέρω βεβαίω ότι η είπατε εκπρόσωπο και οι συνεργάτε τη, ε, όπω είπαμε και χθε, κάνουν θαυμάσια δουλειά. Όπω είδαμε σε σχέση με το Ιράν, είναι λαμπρό ευρωπαϊκό κατόρθωμα. Είναι θαυμάσιο το ότι είπατε εκπρόσωπο και οι συνεργάτε τη έκαναν αυτήν τη θαυμάσια δουλειά και όλοι και εσείς ε, David κάνετε θαυμάσια δουλειά αλλά θα θέλαμε να έχετε λίγο περισσότερη φιλοδοξία, να είστε πιο φιλόδοξοι. Ο David ή ο, ο παρακαθήμενος με την άδειά σας, ε, Πρόεδρε, να πω και εγώ δύο λόγια. Θα θέλαμε και εμείς να σχολιάσουμε. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία αυτή που μας δίδεται για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Το εκτιμούμε ιδιαίτερος πραγματικά, με πάσα ειλικρίνεια. Εκτιμούμε την υποστήριξη και τη δέσμευση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την εκκίνηση της υπηρεσίας αυτής που δεν ήταν απλή, ξέρετε, δεν ήταν μικρό πράγμα. Αυτό που αντιμετώπισε η κυρία Άστον τον πρώτο χρόνο της θετία της ε, ουσιαστικά ε, πρέπει να αντιπραγματευτεί και την νομική βάση και την υπηρεσία που θα την υποστηρίζει. Και με προσπάθησε να δημιουργήσει αυτές τις δομές. Προσπαθούσε και να πετάει το αεροπλάνο όπως ε, λέει και αυτή η χαρακτηριστικά και παράλληλα να χτίζει, να φτιάχνει τα φτερά και τον κινητήρα. Πολλά έχει πετύχει όμω και στο επίπεδο της πολιτική. Το Ιράν αποτελεί ένα τελευταίο παράδειγμα και μόνο. Η κάθε παρουσίασε την αναθεώρηση όπως ζητήθηκε πριν από το καλοκαίρι και εσείς πρόεδρε αναφερθήκατε σε διάφορες περιστάσεις στην χρονική συγκυρία σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν κάπως πρόημη υπό την έννοια ότι κατέληξε στα γραφεία του κόσμου τη στιγμή που ε, εξετάζαμε τις θεσμικές αλλαγές του επόμενου έτους. Ε, έχουμε ευρωεκλογέ, έχουμε εκλογές της Επιτροπή, μετά είναι περίεργη η χρονική συγκυρία και ένα θέμα που απασχολούσε όλους κατά την προετοιμασία της έκθεσης αυτής της αναθεώρησης είναι κατά πόσο θα γίνει η νομική αλλαγή πριν τη θεσμική αλλαγή ή μετά. Νομίζω ότι τελικά τι επικρατεί ως κοινή θέση, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα χρονική στιγμή να ξεκινήσει αυτή η νομική μετατροπή και άρα αναπόφευκτα αξιολογούμε τις διάφορες προτάσεις ε, υπό το φως αυτό στην παρούσα στιγμή για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα ήθελα να αναγνωρίσω την Ηράκλεια προσπάθεια που έχει κάνει η Προεδρία η Λιθουανική και ο πρέσβης έχει αφιερώσει τέσσερις γύρους ανταλλαχών συζητήσεων στα πλαίσια του Κορεπέρ και αυτό και για την προετοιμασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που ελπίζουμε να, να εγκριθούν το Δεκέμβριο από το Συμβουλίο Γενικών Υποθέσεων. Το θέμα ασφαλώς αποτελεί ένα μείγμα διαφόρων στοιχείων σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της ΥΠΑ της εκπροσώπου για την βελτίωση της ε, παραγωγικότητάς μας και στοιχεία τα οποία είναι πιο μεσοπρόθεσμα και τα οποία προαπαιτούν αλλαγές. Αν όχι απαραίτητα της απόφασης για τη σύσταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, αλλά των μεμονωμένων αποφάσεων, των μεμονωμένων κανονισμών. Και ξέρουμε τι συνεπάγεται η αλλαγή, για παράδειγμα, του καταστατικού, του προσωπικού. Αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε τι θα θέλαμε να κάνουμε σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Κάποιες από τις συστάσεις ως σκοπό έχουν να καταστήσουν την αντιπροσωπεία μας πιο παραγωγική. να περάσουν δηλαδή κάποιες οδηγίες στους επικεφαλείς ε, σε ό,τι αφορά και τους προϋπολογισμούς, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τους πόρους των αντιπροσωπιών και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας επιτόπου μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πρεσβειών των κρατών μελών. Εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη δουλειά στο μέλλον σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, ε, μίσθωση από κοινού, εικόνα ευρωπαϊκής ιστορίας κτλ. κτλ. Αυτά σε μέσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν μπορεί να γίνει αυτό άμεσα. Για κάποια στοιχεία τα οποία ήδη θίξατε, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τους δικούς απεσταλμένους. Εδώ θα χρειαστεί μια ξεχωριστή συζήτηση και πιο πολλή χρόνο συζήτησης με τα κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά την Προεδρία των ε, Ομάδων Εργασίας. Εδώ θα χρειαστούμε πολύ χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κάποιων βραχυπρόθεσμων σχεδίων, θα τα κοιτάξουμε αυτά υπό τη δική μας αρμοδιότητα. Ένα δεύτερο τμήμα συστάσεων έχει να κάνει με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, όπως για παράδειγμα η επερχόμενη διαθεσμική μετάβαση σε ό,τι αφορά την ανάθεση των φακέλων, την ιστορική διαρρύθμιση και οργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα σημαίνει ίσως και νομοθετικές αλλαγές. Και αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Αυτό απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς ε, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις φυσικές, ε, φυσικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει και στην εργασία της η ε, υπατή η αντιπρόεδρος, η πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα μπορούσε να ε, ιδρυθεί μια μόνιμη αντιπροεδρία η οποία θα αντιμετωπίζει τα θέματα ad hoc. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε ως ιδέα σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση των θέσεων, των υψηλόβαθμων θέσεων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσεως, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ε, διευθυντών. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει ασφαλώς η διάδοχος ή ο διάδοχος της κάθε Άστον, Πιέρ Βιμόντ, αναφέρθηκε μιλούσα ως Πιέρ Βιμόντ, αλλά είναι αλήθεια και εγώ και ο Πιέρ Βιμόντ έχουμε παίξει διάφορους ρόλους τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι και οι δύο είχαμε την αίσθηση ότι αυτό ήταν σωστό στην φάση της εκκίνησης, όπου ήταν τεράστιες οι προκλήσεις και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ένας μόνο γενικός γραμματέας από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά το προτείναμε και στην κάθε άστον ότι αυτή η σχέση, αυτή η διαμόρφωση δεν χρειάζεται να συνεχίσει στην επόμενη φάση και αυτός ο τετός ρόλος μπορεί να ε, εκτελεστεί από ένα άτομο. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό η μοναδική μεταρρύθμιση που προβλέπετε. Δυστυχώς, όπως είπατε, Πρόεδρε, εξ αρχής, ο Πιέρ σκόπευε να παραβρεθεί. Δεν ήταν στην σύνοδο του Βίλνιου, αλλά δυστυχώς είχε πιο πιεστικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή. Και αυτό, λοιπόν, ε, ε, τον εμπόδισε γιατί έπρεπε να συμμετάσχει σε μια βιντεοδιάσκεψη και δεν μπορούσε έτσι να έρθει στο Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το CSDP, την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία, ασφαλώ είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και σε ό,τι αφορά τι δομέ αντιμετώπιση τη κρίση. Το υφιστάμενο σύστημα μα κάνει να αναρωτιόμαστε σε ό,τι αφορά κυρίω θέματα αναφορά και εκθέσεων, σε ό,τι αφορά επίση τι ευθύνε στα πλαίσια τη ΚΕΠΑ. Αυτό θα σήμαινε όμω αλλαγή θα σήμαινε τροποποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο συντονισμό βέβαια. Αλλά να δούμε καταρχάς τι θα, α, πώς θα εξελιχθούν και οι συζητήσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, του ολοκληρώσουμε την πρότασή μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βρισκόμαστε στην παρούσα φάση, Πρόεδρα. Είπατε κι εσείς ότι χρειαζόμαστε μία αποστολή. Εγώ με πάσα ειλικρίνεια να σας πω, δεν είναι θέμα μάλλον συγγνώμη φιλοδοξίας πρέπει να βρούμε τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα δίλημα κατά πόσον αυτή τη δικασία θα ξεκινήσει τώρα, ξέροντας ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε από θεσμική άποψη προτού αλλάξει η θετία του Κοινοβουλίου και επίσης αναγνωρίζοντας ότι με πάσα ειλικρινία κάποια από τα θέματα αυτά προαπαιτούν και συμμετοχή του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίσης ε, και του Αντιπροέδρου κτλ. Άρα, το δίλημα είναι πραγματικό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τώρα, εδώ και τώρα, κάτι ιδιαίτερα φιλόδοξο, το οποίο δεν θα ολοκληρωθεί ενδεχομένω, ή να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι, κοιτάξτε, θα καταγράψουμε πώς έχει κατάσταση σήμερα και αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν οι νέοι θεσμικοί φορείς όταν θα τοποθετηθούν μετά τις ευρωεκλογέ, μετά την αλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη στην παρούσα φάση δεν θέλουν να ξεκινήσουν μια νομοθετική αναθεώρηση. Προτιμούν απλά να καταγράψουν πώς έχει η κατάσταση και αυτά να τα προωθήσουν στη φάση μετά τις ευρωεκλογέ και μετά το διορισμό της νέας επιτροπής. Αυτά θα ήθελα όμως να πω μόνο στην παρούσα χρονική φάση από πλευρά υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ασφαλώς ο πρέσβης θα μας παρουσιάσει τη δική του άποψη για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Καλύψατε τα περισσότερα θέματα ουσίας. Αυτά θα ήθελα κι εγώ. Καταρχάς, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα αποδώσει πολύ σημασία και μεγάλη προτεραιότητα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και το δεύτερο τμήμα της αναθεώρησης θα γίνει από τη Νέα Επιτροπή και πιθανώς νέο είπα το εκπρόσωπο και φυσικά και ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές. Ο Ντέβιντ ε, εξήγησε γιατί είναι σκόπιμο αυτό Έχουμε αποδεχθεί εμείς ε, αυτή τη συλλογιστική. Και πιστεύουμε ότι ναι μεν υπάρχουν ελλείψεις ε, και αδυναμίες και γι' αυτό δεν είναι εύκολες οι αλλαγές, θέλουμε περισσότερο χρόνο και εξέταση. κατά την προετοιμασία για την Προεδρία μας πριν από δύο χρόνια αρχίσαμε να το συζητούμε πριν από 1,5 χρόνο μας ρώτησαν τότε τι θα κάνουμε με αυτήν την επανεξέταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και η απάντησή μας ήταν πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση και μετά να επανεξετάσουμε τη λειτουργία της είναι πρόσφατος οργανισμός και έχουν γίνει αλλαγές ε, στην νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι πολλά μπορούν να γίνουν χωρίς σημαντικές αλλαγές, να γίνει πιο αποδοτική η διαχείριση, να υπάρξει περισσότερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των αντιπροσωπιών και των πρέσβειών των κρατών μελών να υπάρχει κοινή υποβολή εκθέσεων Τώρα, επί της διαδικασίας, το Κορεπέρ συζήτησε για τέσσερις ομάδες βράχυπρόθεσμων ε, συστάσεων. Πρώτο, λειτουργία της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, που κάτι που έχει να κάνει με τη γενική λειτουργία δηλαδή, αυτό που γίνεται δηλαδή κυρίως από τις Βρυξέλλες. Μετά, εξωτερική εκπροσώπηση, αντιπροσωπείες, πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση για αυτές τις εξωτερικές εκπροσωπήσεις. Το ανέφερε και ο Ντέιβιτ. Συνεργασία με τις πρεσβείες. Κοινή υποβολή εκθέσεων, αλλά και διοικητική απλούστευση. Αυτό μπορεί να γίνει και με τον υπάρχοντα δημοσιονομικό κανονισμό Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει πιο στενή συνεργασία υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και επιτροπής. Τρίτο θέμα. Συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πολύ σημαντικό θέμα. Και εδώ είναι και το θέμα της τελέχωσης. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλλά θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά ικανοποιητική. Αυτή η ποσόστοση τουλάχιστον ένα τρίτο από τις εθνικές διοικήσεις. Βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα πώς εφαρμόζεται, αλλά τονίστηκε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί αυτή η ποσόστοση, αυτή η προσέγγιση. γιατί αυτό σημαίνει κοινή ιδιοκτησία της λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και ε, επίσης θα σήμαινε ότι βασίζεται στην ευρωπαϊκή διπλωματική κουλτούρα και ο τέταρτος πυλώνας ήταν οικονομικά και θέματα προσωπικού. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Συζητήσαμε και για την μακροπρόθεσμη διαχείριση Έχουμε και πιο μακροπρόθεσμα λοιπόν συστάσεις. Είναι πιο θεωρητικές ας πούμε. Η κυριότερη θα έλεγα είναι ότι χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις για τους αναπληρωτές του υπάτου εκπροσώπου. Για το θέμα αυτό όμως ε, το Κορεπέρ ε, θεωρούν, θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική ρύθμιση που υπάρχει τώρα, ότι εκπροσωπείται ο ύπατος εκπρόσωπος από υπουργούς ή από επιτρόπους. Αλλά πιστεύω ότι και αυτό το θέμα θα εξεταστεί ε, στο εγγύς μέλλον. Βεβαίως θέλουμε να υπάρξει βελτίωση αλλά υπάρχει και το θέμα των προξενικών υπηρεσιών. Θα θέλαμε για το θέμα αυτό να υπάρξει μία μικρή έστω βελτίωση. Θα θέλαμε δηλαδή σε καταστάσεις κρίσεων και την προετοιμασία σχεδίων για τα απρόβλεπτα να συμμετέχουν και οι προξενικές υπηρεσίες. Αλλά υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις κυρίως από τα νέα κράτη-μέλη. Ε, έχει πολιτική φύση όμως το θέμα αυτό. Τι άλλα βήματα. Έχουμε λοιπόν ε, τα αποτελέσματα τα πορίσματα του Συμβουλίου, θα τα ξαναδεί η Κορεπέρ και περιμένουμε στις 17 να τα ξαναδεί το Συμβούλιο. Γιατί το πόσο φιλόδοξοι πρέπει να είμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υψηλές φιλοδοξίες. Και τώρα που θα έχουμε νέο κοινοβούλιο, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μάλλον ε, και νέο ύπατο εκπρόσωπο. Οπότε όλα αυτά θα μας επιτρέψουν ε, να κάνουμε δεχομένως και αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε πρώτα επί της ουσίας και θέλουμε και μια επίσημη πρόταση από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Για το θέμα επίσης της Προεδρίας των Ομάδων Εργασίας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μεταξύ κρατών μελών χρειάζονται περισσότερες συζητήσεις σε βάθος ε, και μία επίσημη πρόταση για να αλλάξουμε την κατάσταση. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου θα έχουμε κάποια συμπεράσματα προς αυτή την κατεύθυνση και ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Κομισιόν θα κάνουν ό,τι πρέπει, αλλά φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Και για να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να σκεφτούμε και τι μπορεί να χρειαστεί να επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα το 2015. Ας δούμε όμως πρώτα ποιες θα είναι οι αποφάσεις και οι απόψεις των κρατών μελών και οι απόψεις των κρατών μελών πώς θα εκφραστούν στο Συμβούλιο της 17ης Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να φτάσω αλλά ήμουν ομιλητή στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που είχε μία διάσκεψη και φαντάζομαι ότι στην εισαγωγή του ο κύριος Μπροκ μίλησε για την αναθεώρηση που δημοσιεύθηκε τέλη Ιουλίου και καλωσόρισε το γεγονός ότι αυτή η έκθεση αντικατοπτρίζει διάφορα θέματα ε, που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα περισσότερα θέματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν σε αυτό το κείμενο. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν γι' αυτό. Αλλά χρήσιμο θα ήταν εγώ να εστιάσω σε δύο θέματα. Καταρχάς, ένα γενικότερο θέμα, το οποίο ανέφερε και ο κ. Σάλιβαν. Πώς θα διασυνδέσουμε, δηλαδή, τα βραχυπρόθεσμα θέματα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει και μπορούν να εφαρμοστούν πάρα αυτά με κάποιες πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε νέο κοινοβούλιο και νέα ύπατη εκπρόσωπο ή νέο ύπατο εκπρόσωπο. Φυσικά, είναι δύσκολο πολιτικά να φανταστούμε μία αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου τώρα σε αυτή τη φάση. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το να αφήσουμε σε ένα νέο ύπατο εκπρόσωπο το καθήκον να ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση και, την, και το να βρει, εν πάση λύσεις στα προβλήματα. Ας δούμε τι μπορούμε ρεαλιστικά να κάνουμε και εμείς βέβαια, αλλά και το επόμενο κοινοβούλιο. Η πρότασή μου λοιπόν ποια θα ήταν. Να προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε τη δουλειά αυτή. Να ξεκινήσουμε τη δουλειά για την επόμενη μεταρρύθμιση. Παρά να πούμε, εντάξει, εμεί θα κάνουμε τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα, α πούμε, του μακροπρόθεσμου στόχου, του αφήνουμε στου επόμενου. Γιατί μετά από πέντε χρόνια εμπειρία που έχουμε την υπηρεσία εξωτερική δράση, η σημερινή ηγεσία θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτόν τον προβληματισμό και θα πρέπει να επηρεάσει και την πιο φιλόδοξη μελλοντική μεταρρύθμιση. Έχει σημασία ποιος συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία την νομοθετική. Και για να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή της απόφασης. Αλλά σε ενθαρρύνουμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια αναζήτησης συνέχειας. Γιατί, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί που κάναν καλή δουλειά αυτά, αυτή την πενταετία να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Επίσης, ας εντοπίσουμε και κάποια πιο κρίσιμα σημεία στο πλαίσιο που ανέφερα ήδη. Γενικά υπάρχει ικανοποίηση για την, τις βασικές, τις αδρές γραμμές της αναθεώρησης που δημοσιεύτηκαν. Και για να αναφερθώ σε κάποιες θα μπορούσα να μιλήσω για τη σύμπτωση απόψεων ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της ΥΠΑ της εκπροσώπω ε, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ούτω ώστε να εφαρμόζεται μια συνεκτική προσέγγιση, συνεπής προσέγγιση. Η αναθεώρηση πάντα δεν συνάδει όμω με αυτό το στόχο. Παραδείγματο χάρη. Υπάρχει έλλειψη, δεν υπάρχουν επαρκείς αρμοδιότητες η εξωτερική διάσταση των κοινωτικών πολιτικών είναι κάπως ελλειπής. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε σε περισσότερους αποσπασμένους ε, εθνικούς υπαλλήλους για να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα. Θα πρέπει να μας βοηθήσει και η ίδια υπηρεσία να αξιοποιήσουμε την πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σωστό να έχουμε υπερβολικά ψηλό αριθμό αποσπασμένων εθνικών υπαλλήλων. Ε, αυτό πάνω το θεωρούσε πρόβλημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δείχνουν και τα δεδομένα. Αντίθετα. Παραδείγματο χάρη θέλουμε ε, επίση κάτι άλλο. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση να δημιουργηθεί μια, στο να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή διπλωματία. Να υπάρχει έτσι μια νοοτροπία ότι ανήκουμε σε μια ομάδα. ένα esprit de corps, μια κοινή νοοτροπία. Κάτι μπορούμε να κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση παραπάνω. Κάτι άλλο σημαντικό επίσης για μας, που δεν, δεν μας ικανοποιεί σε αυτό το κείμενο, και υπήρχε και τροπολογία σχετική. Ε, για μία μεταφορά κονδυλίων προς τον, προς τον προπολογισμό της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ένας αυτόνομος προϋπολογισμός. Ε, γιατί τώρα αποτελεί γραμμή του προϋπολογισμού της ΚΠΑ. Θέλουμε να είναι αυτόνομος ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και κάτι πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος. Το θέμα της ε, δημοκρατικής λογοδοσίας, η εφαρμογή του άρθρου 26, σχέση με το Κοινοβούλιο, η δήλωση για την ε, δημοκρατική λογοδοσία. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι αυτό το σημείο λαμβάνεται υπόψη, αλλά πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του βαθμού ε, λογοδοσίας, ούτως ώστε να συνάδει με το ρόλο της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης και με το ρόλο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα. Ε, μία εκ των προτέρων διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εντολές, για τις αποστολές υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε πάρα αυτά. Γιατί μπορεί να γίνει χωρίς καμία νομοθετική αλλαγή. Αυτές είναι οι βασικές μου απόψεις, τα βασικά σημεία που ήθελα να σταθώ και εν κατακλείδη θέλω να πω το εξής. Κάτι που δεν είναι πολύ επίκαιρο, αλλά συνδέεται. Ίσως πρέπει να δείξουμε και κάποια ικανοποίηση. Ε, να είμαστε περήφανοι για την ε, υπηρεσία εξωτερική δράση, για να δούμε τη Σερβία, το Κοσφοπέδιο, ε, το ρόλο που έπαιξε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ήταν πολύ καλός. Μερικές φορές δεν το αναγνωρίζουν αυτό οι εφημερίδες. Αλλά αυτό δεν πρέπει να να μας αποτρέπει από το να αισθανθούμε και αυτή την υπερηφάνεια. Μετά από κάποια χρόνια μπορούμε να αναγνωρίζουμε ότι μετά αρχίζει τέλος πάντων η υπηρεσία αυτή να γίνεται έτσι, πηγή α, πρωτοβουλειών για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Σάλιβαν. Ευχαριστώ και τον κύριο Πρέσβη για τις ε, παρουσιάσεις τους. Θα είμαι ειλικρινής. Εντελώς. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο μέσω της έκθεσης Μπροκ ζήτησε η υπηρεσία αυτή να είναι τμήμα της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έγινε αυτό. Και το Κοινοβούλιο παρόλα αυτά έπαιξε το παιχνίδι όπως έπρεπε. Στήριξε, στήριξε με, πολύ σωστό τρόπο και για τον προϋπολογισμό και για τις προοπτικές και για τον πρώτο, από τον πρώτο χρόνο υποστηρίξαμε τις πιστός πληρωμών, υποστηρίξαμε την ειδική γραμμή για τους ειδικού εκπροσώπους. Δυστυχώς για ένα θέμα νομικής βάσης δεν ε, προχώρησε αυτό. Δώσαμε απαλλαγή το πρώτο χρόνο. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά γιατί η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ήταν θετικό και συμφωνώ με τον απολογισμό που έκανε ο κ. Γουατιέρη ότι χωρίς να κρύβουμε ούτε το καλό ούτε το κακό, αυτό που έγινε αξίζει τα πρώτα αυτά χρόνια. Αλλά καλά τώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, απαλλαγή. Κατά την απαλλαγή, κύριε Σάλιβαν, μέσω του ψηφίσματος πέρα από την Ολομέλεια ζητήσαμε κάτι το λογικό. Δηλαδή να ανοίξει μία αντιπροσωπεία στον Παναμά. Παράδειγμα. Γιατί ο Παναμάς, ε, ο Παναμάς έχει γίνει σημαντική ε, εμπορική και οικονομική βάση. Και δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτήν την αντιπροσωπεία. Συζητάμε κύριο Σάλεμα αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα δημοσιονομικά μέσα. Τα, ξέρετε ότι συζητάμε το μηχανισμό συναπόφασης του, για τη χρηματοδότηση και η Κομισιόν αποφάσισε να αποσύρει τις προτάσεις της για 90 ε, ε, εργαζόμενους στη Λατινική Αμερική. Δεν είναι σοβαρά αυτά, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω, νομίζω ότι όλες οι αντιπροσωπείες της Ένωσης λειτουργούν αποτελεσματικά, ικανοποιητικά. Η τελευταία επίσκεψη που κάναμε στη Washington εμείς ως, ε, ως Επιτροπή και στη Νέα Υόρκη ε, μας πλαισίωσαν υποδειγματικά οι πάλι μας εκεί. Επιμένω, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Γκουαλτιέρη, ότι υπάρχουν αντιπροσωπείες που ακόμη δεν έχουν καταλάβει ότι εκπροσωπούν όλα τα όργανα της Ένωσης. Πρόσφατα έγινε μια επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου μας στην ε, συνάντηση κορυφής των Άνδεων, όπου κάποιος εκπρόσωπος ε, από την ε, αντιπροσωπεία μας εκεί έκανε δηλώσει στον τύπο κατά τον απόψεων του Κοινοβουλίου για συζητήσει που δεν είχαν ακόμη καταλήξει. Θα πρέπει να καταλάβουν οι υπεύθυνοι των αντιπροσωπιών ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα τη Ένωση. Και δεν είναι δυνατόν ένα υπάλληλο να εκφράζεται υπέρ ενό θεσμικού οργάνου και κατά ενό άλλου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με βάση τι συνθήκε βέβαια. Αυτή δεν είναι η γενική τάση. Στι περισσότερε περιπτώσει είναι καλά τα πράγματα και πρέπει να συγχαρούμε του υπευθύνου και ιδιαίτερα τον κύριο Σάλιβαν. Γιατί πέρα από τις άλλες σημαντικές του ευθύνες ε, που αναφέραν προηγουμένως, έχει και την κύρια ευθύνη για την ε, λειτουργία της υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης που από πλευράς διοικητικής και οργανωτικής πάει πολύ καλά. Αλλά είδαμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, θα πάμε καλύτερα. Νομίζω ότι η και εκπρόσωπος είδε τις Απόψη του Κοινοβουλίου και τις έλαβε υπόψη αρκετά τις ε, προτάσεις λοιπόν Μπροκ και Γουαλτιέρη, αλλά το θέμα αυτό δεν το αποφασίζει μόνο η είπατε εκπρόσωπος και λοιπόν τα κράτη-μέλη. Και εδώ τίθεται θέμα. Δηλαδή, να δούμε εάν όλη αυτή η συγκεντρωμένη εμπειρία θα επιτρέψει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα αποφάσεις για να ανταποκριθούμε σε ορισμένες ε, πλευρές που ακόμη δεν είναι ικανοποιητικές. Και επίσης έχει δίκιο ο κύριος Σάλιβαν που λέει ότι θέλουμε να βελτιωθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και είναι καλό πριν πάρουμε αποφάσεις να αναλάβουν οι νέοι αρμόδιοι. Αλλά κάποιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν ε, βράχη πρόθεσμα για να υπάρξουν βελτιώσεις και θα ήταν κρίμα ενώ έχουμε τόση πείρα ενώ έχει συγκεντρώσει τόση πείρα και είπατε εκπρόσωπο και οι συνεργάτε τη, να μην μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτή η πείρα. Υπάρχουν και άλλε υποθέσει. Το ανέφερε ο πρόεδρο ε, το θέμα των προαγωγών. Είναι σημαντικό να υποφεληθούμε από την πείρα των εθνικών διπλωματών, αλλά δεν μπορούμε να αποθαρρύνουμε και τους δικούς μας υπαλλήλους των οργάνων της Ένωσης. Και κύριο Σάλιβαν, θα υπήρχε δυνατότητα και υπάλληλοι του Κοινοβουλίου να περάσουν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό θα βοηθούσε να συμπληρώσετε την οπτική σας, ε, το οπτικό σας πανόραμα. Και καταλήγω λέγοντας ότι είναι σημαντικό και ουσιώδες το Κοινοβούλιο που επετέλεσε τις υποχρεώσεις του έναντι της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης με πολύ ικανοποιητικό τρόπο και με πολύ υπεύθυνο τρόπο στηρίξαμε την ύπατη εκπρόσωπο συμπεριφερθήκαμε με ιδιαίτερα υπεύθυνο τρόπο ε, σε σχέση με τις άτυπες ακροάσεις ε, που κάναμε με τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών. Δεν επικρίναμε κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και από πλευράς οργανωτικής πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που έκανε και η εκπρόσωπος, οι συνεργάτες της οι άλλοι υψηλά ιστάμενοι και ο κύριος Σάλιβαν, ο οποίος είναι οπωσδήποτε μια προσωπικότητα την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε και να τη συγχαρούμε που πετύχαμε αυτό το θαύμα, ότι μπόρεσε να λειτουργήσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό μας ενθαρρύνει και είμαστε σίγουροι ότι σιγά σιγά θα εδραιωθεί αυτή η υπηρεσία και θα μπορέσει να παίξει το ρόλο που του αρμόζει, ούτω ώστε η πολιτική ε, ε, η πολιτική μας των εξωτερικών και της ασφάλειας να είναι πιο αποτελεσματική. Ε, Σας ευχαριστώ συνάδελφοι να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση. Έλαβα ένα email από το Κίεβο μόλις που ότι το αεροπλάνο του Κεντραβιστίσκο 10 μέτρα πριν από την εκκίνηση σταμάτησε, αποφεύχθηκε μία σύγκρουση και έτσι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ε, συνεδρίαση των ε, αρχηγών της αντιπολίτευσης. Αυτό αναφέρθηκε και μέσω Twitter. Πρόκειται για δηλώσεις από την ιστοσελίδα του. Η αυτοκρατορία αντιπιτίθεται, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κρόνμπεργκ. Thank you, Chairman. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να, ευχαριστη... να σας ευχαριστήσω για τις απόψεις σας. Είμαστε περήφανοι για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και για την ε, Συμφωνία Σερβία-Κοσφοπέδιο και σε ό,τι αφορά την πρώτο βήμα για την Συμφωνία με το Ιράν. Δύο ερωτήσεις να κάνω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό πάντα αποτελούσε θέμα συζήτησης ε, σε ό,τι αφορά τη δομή της οργάνωσης. Πείτε μας την άποψή σας η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, να υπάρχει πιο συνεκτική προσέγγιση. Δεύτερη ερώτηση για το Ιράν και νομίζω ότι πολλές φωνές ε, ζητούν αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν. Έναν ειδικό απεσταλμένο τώρα που θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Πείτε μας λοιπόν την απόψη της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η δική μου η ομάδα πάντα ήταν αντιστακτική και επιφυλακτική για το ρόλο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και για το κατά πόσο χρειαζόταν καν. Και θεωρούμε ότι ήταν μια sui ε, υπηρεσία με τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και με καθοδήγηση ουσιαστικά μιας διακυβερνητικής ατζέντα με κάποιο βαθμό δημοκρατικού ελέγχου. Αλλά παραμένουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ο ρόλος, για παράδειγμα, των αντιπροέδρων, των υφιστάμενων η κάθε δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι ενδεχομένως χρειάζονται κάποιοι αναπληρωτές υπό ε, ε, τη εκπρόσωπη σε ό,τι αφορά επίσης ε, το γεωγραφικό τρόπο διορισμού των ατόμων αυτών, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί αντιπροσωπιών και πρώην και ακαδημαϊκοί. Πρόκειται για μια υπηρεσία υπό την καταθήγηση δημοσίων υπαλλήλων και το όλο θέμα που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Βαλκάνια, τη διεύρυνση κτλ. Ποιος είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο. Αυτά λοιπόν είναι απάντητα ερωτήματα. Ήμουν πιο πολύ διστακτικός και επιφυλακτικός. Είμαι κάπως λιγότερο πρέπει να ομολογήσω μετά από τέσσερα χρόνια. Μετά από την εκπληκτική δουλειά που έκαναν και μετά από μια τεράστια κρίση και στην Ευρωζώνη κτλ. Σύστησαν και εδραίωσαν μια υπηρεσία από το μηδέν, από το πουθενά. Τεράστιο επίτευγμα. Σύμφωνο όμως με τον συνάδελφο Σαλαφράγκα, υπάρχουν ε, ιστορικές κληρονομιές σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, αποστολές ε, που δεν υπάρχουν στον Παναμά, στην Κεντρική Αμερική. Και θα θέλαμε να υπάρχει και αποστολή στο Μπαρμπέιντος, ε, όπου φαντάζομαι ότι το κίνητρο των κοκτέιλ στην παραλία είναι πολύ μεγάλο. Πιστεύω, όπως είπαν και οι πράσινοι συνάδελφοι, θέματα όπως η Πρίστινα, το Κωσυφοπαίδιο, οι συζητήσεις με το Ιράν, αποτέλεσαν σημαντικά επιτεύγματα για τη Βαρόνη Άστον και για την υπηρεσία. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Το συζητήσαμε και πριν από κάποια χρόνια όταν επισκεφτήκατε το γραφείο μου. Θα πρέπει να δούμε πιο πολλά παραδείγματα προς τη αξίας που γλιτώνουν χρήματα ιδιαίτερα των εθνικών προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, την ε, από κοινού εκμίσθωση γραφείων, όπως για παράδειγμα στο Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν. Τέτοια παραδείγματα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα από πολιτικής άποψης ε, και εξηγούν γιατί χρειάζεται μια τέτοια υπηρεσία και οι προξενικές ε, υπηρεσίες. Μπορεί να μην τον υποστηρίζουμε εμείς από πλευράς της ομάδας μου, αλλά ίσως για μικρές χώρες, ίσως αυτό να είναι ένα επιχείρημα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στο εκλογικό μας ε, κοινό. Γιατί δάλλως θεωρώ ότι δεν είναι αμφισβητήσιμη η αξία μάλλον του project. Ευχαριστώ, θα πρέπει να φύγει ο πρέσβης για να προλάβει και τον Πρωθυπουργό που είναι εδώ σήμερα. Και γι' αυτό λοιπόν θα του δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει τώρα και μετά θα ακούσουμε τον Ντέιβιντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τις απόψεις ε, του Συμβουλίου και της Κορεπέρη. Αν μου επιτρέψετε, θα ξεκινήσω από πλευρά ε, Συμβουλίου για να σας απαντήσω. Όντως και πάλι πιστεύω ότι είμαστε υπέρ της ε, φιλοδοξίας ε, του έργου της Υπηρεσίας της Δράσης και της ενίσχυσης της σημαντικής αυτής θεσμικής υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την πολιτική, την εξωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε ο κ. Γκαλτιέρη σε θέματα συνέχειας. Υπάρχει σαφώς συνέχεια μεταξύ του βραχυπρόθεσμου και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου. Αν διατρέξουμε τον κατάλογο των συγκεκριμένων ερωτημάτων. Να σας πω για παράδειγμα οι βελτιώσεις στον τομέα της ενοποιημένης προσέγγισης, της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο στόχο αποτελεί αυτό. Υπάρχει πραγματικά συνέχεια εναρμόνιση του προγραμματισμού και σε ό,τι αφορά το συντονισμό με τις αποστολές και ΕΠΑ. Υπάρχουν διάφορα θέματα, ο ρόλος της Επιτροπής και της υπατής εκπροσώπου. Και εδώ υπάρχει η βραχυπρόθεσμη προοπτική για την είπατη εκπρόσωπο στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και σε ό,τι αφορά τον επικεφαλής της ε, Επιτροπής την ομάδα Relex. Τα συζητάμε εδώ αυτά, αλλά είναι σαφή για το μέλλον. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα αυτό της συνέχειας έχει να κάνει και με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των αντιπροσωπιών. Σας είπα λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να περιορίσουμε το διοικητικό κόστος σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες αυτές και σε ό,τι αφορά και το δημοσιονομικό κανονισμό. Επίσης, ε, για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που ακούσαμε σε ό,τι αφορά την μεταφορά, για παράδειγμα, των εθνικών διπλωματών και γενικά του, προσωπικού, του διπλωματικού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο χρειάζεται στοιχεία και είναι τουλάχιστον απαραίτητο να διατηρήσει αυτό το 1 τρίτο, το ποσοστό ενό τρίτου από τα εθνικά κρατημέλη. Οι κυβερνήσει το συζητούν επισταμμένο στο θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν αυτέ οι διπλωματικέ δυνάμει τη Ένωση. και αφενός, αφετέρου καταλαβαίνουμε βέβαια ότι απαραίτητο είναι να υπάρχει και συνέχεια. Το 1 τρίτο δεν αποτελεί όριο, αλλά είναι απαραίτητο ποσοστό για να υπάρξει συνέχεια αυτή που επιθυμούμε. Σε ό,τι αφορά και τους θεσμικούς αντιπρόσωπους που χρειάζονται, σε ό,τι αφορά νομικά, θεσμικά θέματα, θα πρέπει να αλλάξει ενδεχομένως η νομική βάση. Σε ό,τι αφορά Κοιτάξτε, έχουν γίνει επίσημες προτάσεις ε, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αλλαγή της γραμμή του προπολογισμού του τομέα του προπολογισμού. Αλλά καταρχάς θα πρέπει να γίνουν σωστέ ε, και καλές συζητήσει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες στον κλάδο αυτό. Σε ό,τι αφορά και το... σε ό,τι αφορά την ε, ισορροπή και σωστή χρήση των πόρων. Συνοψίζοντας, ενδεχομένω να επαναλάβω αυτά που είπα, αλλά να πω ότι ναι, το Συμβούλιο είναι υπέρ μιας ισχυρή υπηρεσία εξωτερική δράση, γιατί αυτό αποτελεί ασφαλώς τη βασική οργάνωση, τη βασική ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν συνηθίζω να παρευρίσκομαι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά η αξιολόγηση που μας παρουσιάστηκε έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και χωρίς να είμαι τακτική εδώ, θέλω να χαιρετήσω και εγώ τη δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που ήμουν είτε σε αντιπροσωπεία του Προέδρου του Κοινοβουλίου ή σε άλλες αντιπροσωπείες σε διάφορες χώρες, βλέπουμε ότι η, η συνεργασία γίνεται και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ούτω ώστε να συνεργαστούμε με τους ντόπιου. Αυτά που μπορούν να βελτιωθούν τώρα, ειδικά για μια περιοχή του κόσμου, τη Μεσόγειο. Υπάρχουν διάφοροι φορείς. Η Ένωση για την Μεσόγειο, που με την εκτελεστική της, τον εκτελεστικό της βραχίωνα και τον νομοθετικό της βραχίωνα εντός αγωγικών, ε, την, ε, τον την κοινοβουλευτική συνέλευση, αυτή δηλαδή η ένεση για την ε, Μεσόγειο και με τις διάφορες task force που έγιναν σε διάφορες χώρες, στην Τινησία, στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο, τις συστάσεις που απέρευσαν από τις ε, εκλογικές ε, αποστολές. Ίσως καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά πέστε μου πώς θα μπορούσαμε σε αυτή την περιοχή να εμπλέξουμε τους διάφορους φορεί φορείς και τις διάφορες πρωτοβουλίες που κάνουν οι μεν και οι δε στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάπως έτσι να τις ομαδοποιήσουμε. Είτε που γίνονται στα πλαίσια των, που γίνονται από, στα πλαίσια των, των παρατηρήσεων εκλογών ή των μεικτών task force ε, κομισιών κοινοβουλίου κτλ. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτές να τις βάλουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να μην έχουμε επικαλύψεις. Πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα, πιο ορθολογικά αν θέλετε, ούτως ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη Μεσόγειο. Ε, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι χώρες αυτές της Μεσογείου περιμένουν πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κατά την άποψή μου η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια και η δράση της Υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης είναι καταστροφική. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα, θα σας θυμίσω τον ολέθριο ρόλο στον πόλεμο της Συρίας και στην εξαγωγή οπλισμού ε, σε αυτή τη χώρα. Θα σας θυμίσω τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική. Θα σας θυμίσω τι γίνεται τώρα με, την, ε, ε με τους γείτονες στην ε, Ανατολική Ευρώπη. Το γεγονός δηλαδή ότι όλο και περισσότερες χώρες δεν θέλουν ιδιαίτερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει και τα διέξοδα αυτής της πολιτικής. Για μένα είναι ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί όπως είπε και ο κύριος Σαλαφράνκα, και το έχει πει και ο κύριος Μπαρόσο, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης και όχι τα συμφέροντα των λαών, τα συμφέροντα της σταθεροποίησης, της σταθερότητας και της ειρήνης. Απόδειξη γι' αυτό είναι το χθεσινό άρθρο στο Der Spiegel που σχολίαζε τα αποτελέσματα της συμφωνίας για το Ιράν λέγοντας ότι οι γερμανικές βιομηχανίες τρίβουν τα χέρια τους για τις μεγάλες εξαγωγές και τις μεγάλες δουλειές που έχουν τώρα στο Ιράν μετά την ε, συμφωνία της Ιρανικής κυβέρνησης. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο κύριο ε, Σόλιβαν με τα ζητήματα αυτά. Ε, είναι σημαντικά αυτά που μας είπατε, αλλά πιστεύω ότι τους ψηφοφόρους και τους εργαζόμενους ενδιαφέρουν πιο ουσιαστικά ζητήματα. Είπατε παραδείγματος χάρη ότι τα κράτη-μέλη τώρα θα περιοριστούν σε μια καταγραφή των απόψεων και θα αφήσουν τις αποφάσεις μετά τις ευρωεκλογέ. Εάν κατάλαβα καλά και αν είναι έτσι, είναι προφανές γιατί συμβαίνει αυτό γιατί θα είναι δυσάρεστες οι αποφάσεις και δεν θέλουν βέβαια να εισπράξουν το δυσάρεστο πριν από τις ευρωεκλογέ. Ε, θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι στη Γερμανική Βουλή έγινε συζήτηση για την επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη και με αφορμή αυτή την τοποθέτηση στη Γερμανική Βουλή μάθαμε ότι υπάρχει έγγραφο της υπηρεσίας σας από τις 18 Απρίλη που αφορά το Conops Plus για την επιχείρηση ε, επιτήρησης των, των συνόρων στη Λιβύη, η οποία, το οποίο ντοκουμέντο είναι απόρριτο. Γιατί είναι απόρριτο κύριε Οσόλιβα. Γιατί είναι απόρριτο ένα ντοκουμέντο που αφορά την επιτήρηση των συνόρων ε, στη Λιβύη. Και ένα δεύτερο, υπάρχει επίσης ένα κείμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, που αφορά το ίδιο θέμα με ημερομηνία 19 του Νοέμβρη που προβλέπει τη λήψη στρατιωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστών ε, όσον αφορά από τη βία από άλλες χώρες. Από πού αντλεί το δικαίωμα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να στρατιωτικοποιεί τα ζητήματα αυτά. Τέλος, θέλω να σας πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο μετατρέπεται σε έναν στρατιωτικό συνασπισμό. Και δεν ξέρω αν έχετε ορισμένε πληροφορίε πού πάμε με τη Σύνοδο Κορφή για την άμυνα που θα γίνει το Δεκέμβρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη ανοχή Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο. Κύριε Μπρόκ, μετά θα τον πάρω. Γνωρίζουμε την θερμή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν προσπαθήσαμε να στήσουμε την υπηρεσία. Ο κ. Σαλαφράνκα ανέφερε διαφορετικού τομεί, ε, διοικητικού και ε, αλλά και το θέμα του προπολογισμού και κυρίως η κάθε εκτιμάει την πολιτική σας υποστήριξη. Και ελπίζω να αισθάνεστε ότι και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ε, ερχόμαστε συνέχεια και, και εγώ και διάφοροι άλλοι υψηλά ιστάμενοι να σας ενημερώ. Ερχόμαστε, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε και να σας εμπλέξουμε στη δουλειά που κάνει η υπηρεσία μας όσο γίνεται. Σας ευχαριστώ επίσης για τα σχόλια που κάνατε για την πρόοδο που σημειώθηκε. Νομίζω ότι όλοι εργαστήκαμε πυρετοδός για να στήσουμε την υπηρεσία. Το προσωπικό και του ζητήσαμε πάρα πολλά να κάνει. Όχι πάντα σε εύκολες συνθήκες, σε περίοδους αλλαγής, ε, ε έγιναν μεταθέσεις από όργανα σε όργανα, ε, άραξαν καριέρα ορισμένοι, ε, διάφοροι προσωρινοί υπάλληλοι από τα κράτη-μέλη ήρθαν στην υπηρεσία μας κτλ. Του ζητήσαμε πολλά. Και ανταποκρίθηκε το προσωπικό. Όλο το προσωπικό τη υπηρεσία εκτορική δράση έδωσε την ψυχή του, α πούμε, αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά κανένα δεν δούλεψε τόσο σκληρά όσο εκάθι. Για τη, Σερβία, το, για τη Σερβία, το κοσφοπέδιο, ξέρετε πώς έκανε. Ε, και αισθάνεται ότι έχει την υποστήριξη μια καλή υπηρεσία, αλλά ξέρετε και τα διπλωματικά, πολιτικά ε, προσόντα της, που την ε, κατέστησαν ικανή να κάνει πολλά πράγματα. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τις σχέσεις μας, ε, να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο, τις πολιτικές σχέσεις με τις χώρες, ε, τις εξελίξεις ε, που υπάρχουν γενικά, ούτως ώστε να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Επίσης, κύριε Αγκουράκη, δεν, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που είπατε, ότι είναι μια στρατιωτικοποιημένη οργάνωση εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Καθόλου τη στρατιωτικοποίηση. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε, χάρη στην υπηρεσία, είναι να συνδέσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο και δημιουργούν τις πολιτικές κρίσεις, ε, θέλουμε να τα λάβουμε υπόψη μας για να υπάρξει μια πρόληψη. Μερικές φορές χρειαζόμαστε και πολιτικά, α, στρατιωτικά α, ε, στοιχεία, στρατιωτικό δυναμικό για να το καταφέρουμε αυτό, να αποτρέψουμε τις κρίσεις. Τώρα, γιατί έχουμε ένα μυστικό έγγραφο για τα σύνορα. Είναι γιατί ίσως είναι ευαίσθητα θέματα, ας πούμε. Είναι ευαίσθητα αυτά τα θέματα, λεπτά και παίζονται ζωές ανθρώπων σε αυτές τις αποστολές. Έχουμε 7.000 ανθρώπους σε πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές. Ο κόσμος ρισκάρει τη ζωή του για να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ένωσης, που είναι η πρόθεση Τη ειρήνη και τη σταθερότητα Δεν είναι η στρατιωτική στόχη, είναι η πρόθεση και η διασφάλιση τη ανθρώπινη ζωή. Και εμεί προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και το είδα αυτό το πράγμα στην πράξη. Μπορέσαμε με τη νέα υπηρεσία και με τον τρόπο που λειτουργεί να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή τη η, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που μπορεί η Κομισιόν, πρόληψη των κρίσεων, ανθρωπιστικέ παρεμβάσει, με στρατιωτική υποστήριξη και ενδεχομένω και στρατιωτική παρέμβαση για να σταθεροποιήσουμε καθεστώτα ή να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να αλλάξουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής όπως έγινε στο Μαλί λοιπά. Ή επικοδομητική προσπάθεια στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας με τη βοήθεια της Κομισιόν. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πει πραγματικά μια καλή ιστορία για το τι γίνεται στη διεθνή κοινότητα. το χάρη η Συρία. Εκεί είναι ένα τομέα όπου δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε την ανθρωπιστική καταστροφή. Αλλά μπορώ να σα πω ταπεινά ότι δεν είναι επειδή δεν το θέλαμε να το κάνουμε ή δεν μπορούσαμε, αλλά γιατί υπάρχουν άλλα εμπόδια που δυστυχώ δεν, δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε. Έχουμε μια πλήρη, μια συνεπή, συνεκτική προσέγγιση που είμαστε στις, στα σπαργανά της ακόμα και έχει, πρέπει να σας πω, τεράστιο δυναμικό, ας πούμε. Μπορούμε να αποτελέσουμε μια δύναμη ε, καλοσύνης και σταθερότητας ε, στην παγκόσμια σκηνή. Τώρα κάποια πιο πεζά θέματα συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, κύριε Τάνοκ. Υπάρχουν εξοικονομήσεις. Ήδη τώρα. Αν κοιτάξουμε την κατάσταση στην Ιεμένη, έχουμε μια πολύ καλή ε, συνεργασία με τις Ισπανικές αρχές, για γνωστούς λόγους δυστυχώς. Μειώνουμε την διπλωματική εκπροσώπηση, φτάνουμε σε μια συμφωνία, όταν κλείνει μια πρεσβεία, ας πούμε, και αν θέλουν, ας πούμε, στην ε, αντιπροσωπεία μα να αφήσουν κάποιον, ας πούμε, Ισπανό διπλωμάτη, αυτό ο άνθρωπο δουλεύει εν μέρη για μα, αλλά λειτουργεί και εξ ονόματο, ας πούμε, της χώρας του, στον εμπορικό, ας πούμε, τομέα. Και στην περίπτωση τη Ιεμένη, γλιτώσαμε, εξοικονομήσαμε 500.000 ευρώ. Τεράστιο όφελο. Είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, το λέω γιατί ξέρετε τι γίνουμε, προσπαθούμε να νοικιάσουμε κτίρια, τι γίνεται με τα νίκια, όταν ανοίγουν και κλείνουν γραφεία υπάρχουν διάφορα οικονομικά θέματα, αλλά πραγματικά τα κοιτάμε όλα αυτά πάρα πολύ σοβαρά. Και σε 5-10 χρόνια πιστεύω ότι θα συστεγαστούμε ακόμα περισσότερο, ε, πρεσβείες και εμείς ας πούμε, ή επίσης ε, πρέσβεις ας πούμε ε, κρατών μελών ε, που δεν εκπροσωπούνται, δηλαδή που δεν βρίσκονται στη χώρα εκεί έρχονται απλώ για μια επίσκεψη. Μπορεί να ενημερωθούν από το προσωπικό μα, να χρησιμοποιήσουν τα γραφεία μα, το, του κομπιούτερ κτλ. Να υποφεληθούν από την υποδομή μα δηλαδή. Και πιστεύω και το θέμα των, προξεν... των προξενείων θα λυθεί σε κάποια φάση. Φυσικά εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Φράση. Δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε αυτό. Αλλά υπάρχουν δυνατότητε συνεργασία εδώ, χρησιμοποιώντα τα κτίρια τη υπηρεσία μα, ούτω ώστε να υπάρχουν κάποιε κοινέ προξενικέ ε, δραστηριότητε. Ούτω ώστε να προωθούμε και τη δράση μας. Επίσης προσοχή όταν λέμε ότι στο, στο, στην κατελα, στο κατελάκι μας, ας πούμε, στην ετικέτα μας, ότι εδώ μπορείτε να χτυπήσετε την πόρτα όσο έχετε προβλήματα και είσαστε Ευρωπαίοι πολίτες, ας πούμε, να υπάρχει κάποιος από πίσω που να μπορεί να το απαντήσει στο, πρόβλημά του και να του το λύσει. Για τη στελέχωση. Εγώ όταν συναντώ έναν άνθρωπο, ε, δεν ξέρω αν είναι αποσπασμένος, αν είναι μόνιμος, αν είναι προσωρινός υπάλληλος κτλ. Εγώ βλέπω μόνο επαγγελματίε, ικανότατου. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Είτε αν κάποιο είναι διπλωμάτη, α πούμε, ενό κράτου μέλου αποσπασμένο, αν είναι κάποιο, πούμε, προσωρινό υπάλληλο αποσπασμένο, ή αν είναι ε, ευρω, ευρωπαϊκό ε, υπάλληλο, α πούμε. Δεν ξέρω αν δουλεύει στην Κομισιόν, αν δουλεύει στην Γραμματεία του Συμβουλίου, δεν έχω ιδέα και δεν νομίζω ότι έχει και σημασία. Και θα ήταν λάθος να πούμε ότι όσοι έρχονται ας πούμε, από τα ξένα υπουργεία Εξωτερικών, ας πούμε, δεν έχουν έτσι, κίνητρα. Αντίθετα, έχουν απίστευτες γνώσεις που δεν τις έχουμε κατά ανάγκη εμείς στην υπηρεσία, τις φέρνουν ας πούμε, και, τις, ε, και μας διαποτίζουν αυτές. Παραδείγματο χάρη, η εξωτερική διάσταση εσωτερικών πολιτικών, ας πούμε, ε, η παραδείγματο χάρη η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική νερού κτλ. Η κινητικότητα, μετανάστευση. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα. Ε, το θέμα δεν είναι να βρούμε τσακ ένα γραφειοκράτη, ένα μολύβο πρόχτη που θα μου γράψει ένα χαρτί. Το θέμα είναι να βρούμε ένα πραγματογνώμονα. Συχνά τα κράτη-μέλη έχουν αυτή την πραγματογνωμοσύνη και φυσικά συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν και ξέρω ότι τελικά η καλύτερη συνεργασία μεταξύ της δικής μας υπηρεσίας και το να λάβουμε υπόψη μας την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών, αυτό μπορούμε να το ξαναδούμε λιγάκι, γιατί εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που λείπουν. Βέβαια, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Η Κομισιόν είναι πάρα πολύ καλή υπηρεσία. Έχουμε βέβαια τις διαφορές μας και πάντα θα τις έχουμε. Αλλά νομίζω ότι βελτιωνόμαστε και εμείς και εκείνη συνέχεια και βοηθάμε την Κομισιόν στο έργο της για, για εσωτερικές πολιτικές που έχουν και μια εξωτερική διάσταση. Για την οργάνωση τώρα. Ποτέ δεν λέει κανείς, α, έχουμε την τέλεια οργάνωση. Συνέχεια βελτιώνεται η οργάνωση και έχω κάποια εμπειρία από την ε, Ευρωπαϊκή Υπαλληλία. Πρέπει συνέχεια να ξαναβλέπεις τα συστήματά σου, τις δομές σου, το οργανόγραμμά σου για να βελτιώνεις τις επιδόσεις σου. Πιστεύω ότι θα υποστεί διαδοχικές μεταρρυθμίσεις, προσαρμογές και αλλαγές οι υπηρεσίες μας. Βέβαια για το θέμα του βραχυπρόθεσμου, παύλα, μακροπρόθεσμου, αυτό είναι και πολιτική επιλογή, έτσι. Επίσης, επειδή σεβόμαστε ε, και τα αποτελέσματα των εκλογών, ε, το διορισμό της νέας Κομισιόν και του νέου ύπα του εκπροσώπου, υπάρχει το θέμα του κατά πόσο θα προδικάσουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα, εάν αποφασίσουμε τώρα. Θα, προδικάσουμε, δηλαδή, σε κάποιο βαθμό, το αποτέλεσμα των εκλογών. Το να εντοπίσουμε τώρα το μενού των θεμάτων που πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθούν, μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να αφήσουμε επαρκή ελευθερία στον επόμενο πρόεδρο και τα λοιπά και είπα το εκπρόσωπο για αυτά τα θέματα. Εσείς θα συζητήσετε και με, τον ένα και με τον άλλο. Πρέπει ούτως ή άλλως να δείτε, ε, να το συζητήσετε, να πείτε τι προσδοκάτε. Πρέπει να βρούμε αυτήν την ισορροπία. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα θα έχουμε όλες τις απαντήσεις. Τελείωσε. Γιατί αυτοί οι νέοι άνθρωποι που θα έρθουν θα έχουν τις δικές τους ιδέες και θα πρέπει να μπορούν να τις εκφράζουν. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι και λυπάμαι αν το έκανα. Για το θέμα των αντιπροσωπιών μας. Ελπίζω να αισθάνεται το Κοινοβούλιο ότι εξυπηρετούμε καλά τα συμφέροντά σας με τις αντιπροσωπείες μας. Θέλουμε να υπηρετούμε σωστά το Κοινοβούλιο για το θέμα των δικτύων. Αν θα πρέπει να ανοίξουμε στον Παναμά ή στην Τεχεράνη κάποια στιγμή, αυτά είναι περίπλοκα θέματα. Γιατί υπάρχουν και περιορισμοί στους πόρους, έτσι, άρα πρέπει να κάνουμε επιλογές, δεν μπορούμε να ανοίξουμε παντού δεν είναι εύκολο να πούμε κλείνουμε αυτή την προσωπία και ανοίγουμε την άλλη. Γιατί όταν κλείνει μια την προσωπία μερικέ φορέ για λίγα λεφτά, επειδή θα πρέπει να δώσει αποζημιώσει, α πούμε, και να, ε, στο προσωπικό κτλ., ε, σου κοστίζει περισσότερο το κλείσιμο. Άρα τα λεφτά που γλιτώνει από το κλείσιμο δεν τα δίνει για το άνοιγμα μια νέα αντιπροσωπεία. Αυτέ οι συζητήσει πρέπει να τι κάνουμε. Έτσι. Σίγουρα. Είμαστε το έκτο μεγαλύτερο διπλωματικό δίκτυο στον κόσμο. Είναι τεράστιο θέμα αυτό το κληρονομήσαμε από την Κομισιόν και νομίζω ότι είναι η βάση τη δουλειά τη υπηρεσία ε, και αυτή τη βάση πρέπει να τη διασφαλίσουμε. Θα πρέπει τώρα να δούμε πώ μπορούμε να επεκταθούμε με δεδομένη τη βάση. Άκουσα και τι υποδείξει σα ε, για το πού θα πρέπει να επεκταθούμε, σε ποια τμήματα του κόσμου που δεν είμαστε τώρα παρόντε. Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να τη συνεχίσουμε. Να σταματήσω, Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχουν σίγουρα θέματα που παρέλειψα και δεν απάντησα, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους τους βουλευτές για τις ενισφορές τους, για τις παρατηρήσεις τους. Εκτιμούμε πάνω από όλα τη σχέση μας με την Επιτροπή σας, την υποστήριξη που μας δείχνετε. Υπό την ηγεσία της κάθε πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει μια ισχυρή υπηρεσία που έχει την ικανότητα να υλοποιήσει τις πολιτικές φιλοδοξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις και ελπίζω αυτή την κληρονομιά να τη διασφαλίσουμε και να τη διαφυλάξουμε. Αλλά ξέρω ότι μπορούμε να την αναπτύξουμε περαιτέρω στο μέλλον. Αυτή η υπηρεσία έχει τεράστιο δυναμικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο μέλλον και θα το υλοποιήσει, το ξέρω. Ελπίζω να της δοθεί ο πολιτικός χώρος και η διοικητική δυνατότητα να μπορέσει να αναπτυχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί το πιο σημαντικό θέμα που θα αντιμετωπίσουμε στον 21ο αιώνα είναι ο ρόλος που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Και ο τρόπος για να το πετύχει αυτό, να πετύχει ένα ισχυρό ρόλο, είναι μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Κύριος Γκουαλτιέρη, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε για μία σειρά θεμάτων και είναι σημαντικό που συμφωνούμε και συμφωνώ επίσης σε ό,τι αφορά την ε, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική σε σχέση με το τρέχον κοινοβούλιο και το επόμενο. Το θέμα είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ συνέχειας και πλήρης αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που υπάρχει και σε ό,τι αφορά και το πολιτικό περιθώριο ε, λιγμών στους νεοεκλεγέντες αξιωματούχους. Θεωρώ όμως ότι θα μπορέσουμε να το χτενίσουμε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Ως επικεφαλής παρατηρητής ε, στο κοσφοπέδιο το ζω αυτό και πρέπει να πω ότι ναι μεν ε, καταλαβαίνω τι κάνει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και καταλαβαίνω όμως ε, σε ό,τι αφορά τις επίσημες διπλωματικές ε, ε, αντιπροσωπείες και τα λοιπά και τους αποσπασμένους. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαφορετικό επίπεδο δέσμευση σίγουρα, αλλά το θέμα είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια. Να μην πισωγυρίζουμε, να μην χάνουμε πόρους όταν δεν δίνουμε κίνητρα στα άτομα αυτά. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι, θεωρώ. Δεν έχω ιδιαίτερα κάτι να προσθέσω. Ο Έλμαρ θέλει να μιλήσει ίσως και να κάνει κάποια καταλητικά σχόλια. Ο κύριος Μπρόκ. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας και τη συζήτηση από εδώ και πέρα και θα δούμε ποιες θα είναι οι επερχόμενες πρωτοβουλίες και τα μελλοντικά βήματα. Ας ελπίσουμε ότι η συζήτηση θα προχωρήσει στην τρέχουσα θητεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, David. Ήταν πραγματικά υπέροχο που είχαμε εδώ μαζί μας ε, όλο το απόγευμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Χαρά μου, λέει ο κύριος Οσάλβαν. Willst du die begrüßen? Die kommen jetzt. So we will start immediately with the Americans. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την αντιπροσωπεία των Αμερικανών. So, ladies and gentlemen, please take your seat. We come to point 16 of our agenda. Exchange of views. Ανταλλαγή απόψεων με τους φίλους μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Κρίστοφα Μέρφυ που είναι πρόεδρος της Υποπιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γερουσίας μαζί του είναι το μέλος Βουλής αντιπροσώπων Διαθ Μπαλάρ, που είναι μέλος ε, της Επιτροπής ε, για τον Διατλαντικό Διάλογο και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Gregory Mix, που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Νομίζω ότι είναι πολύ σκόπιμη η στιγμή που έχουμε αυτή την επίσκεψη από τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ. Η Επιτροπή μα έχει συζητήσει τι τελευταίε εβδομάδε μαζί με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών τρόπου για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην διατλαντική εταιρική σχέση μετά τι αποκαλύψει για μαζική ηλεκτρονική επιτήρηση από την ε, Υπηρεσία εθνική ασφάλεια και ορισμένε ευρωπαϊκέ ε, υπηρεσίε πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επανέλθει η εμπιστοσύνη γιατί θέλουμε να εμβαθύνουμε τις διατλαντικές σχέσεις. Χρειαζόμαστε αυτή την συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και έχουμε οικονομικά και εξωτερικά συμφέροντα κοινά που θα πρέπει να μας επιτρέψουν να έχουμε επιτυχείς διαπραγματεύσεις για τον διατλαντικό διάλογο και για την συμφωνία για το εμπόριο και, τα, και τις επενδύσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα να μας επιτρέψουν να ε, υπερβούμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τρία ζητήματα σε σχέση με αυτό. Πρώτον είναι η συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, πώς μπορούμε να στοχεύσουμε αυτή τη συνεργασία και όχι να κατασκοπεύουμε τους πάντες. Και τρίτον, ένα θέμα που προηγείται. Πώς θα προστατεύσουμε την ιδιωτική σφαίρα των πολιτών μας δηλαδή προστασία των ιδιωτικών στοιχείων, των δεδομένων, η συμφωνία πλαίσιο, η συμφωνία ομπρέλα για την προστασία των δεδομένων που διαπραγματεύτηκε η κυρία Ρέντινγκ στην Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα και είχατε μια συνάντηση σήμερα ε, με την κυρία Ρέντινγκ και η συμφωνία, του, το θέμα μάλλον του ασφαλούς καταφυγίου και το θέμα της ε, συνεργασίας για το θέμα αυτό πιστεύω και αυτή ήταν εντύπωση που αποκόμισα πριν από τέσσερι εβδομάδε στην επίσκεψη στη Washington με την προσωπία τη ΑΦΕΟ, ότι υπάρχει ζήτηση για το θέμα αυτό εντό των Πολιτειών και ε, κύριε Γερουσιαστά και μέλη τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ξέρω ότι σα ενδιαφέρει αυτό. Και βεβαίω είναι διαφορετικέ οι σχέσει μα ε, με εσά από ότι με τη Ρωσία και την Κίνα, διότι η δημοκρατία και το κράτο δικαίου λειτουργεί στι ΗΠΑ και γίνεται διάλογο για τα θέματα αυτά. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τι σχέσει με άλλε χώρε Γι' αυτό οι φίλοι μα στο Κογκρέσο είναι όντω φίλοι μα. Είμαστε κοινοβούλοι από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού και πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ιδιωτική σφαίρα και ασφάλεια. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτή είναι και ήταν πάντα η ευθύνη των κοινοβουλίων. Και θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι. Βεβαίω μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάθε λεπτομέρεια, να νωρί ακόμη γι' αυτό, αλλά η βούληση να το συζητήσουμε για να επιτύχουμε αυτή τη σωστή ισορροπία για να επανέλθει η ε, εμπιστοσύνη και να προωθήσουμε το θέμα της συμφωνίας TTIP που δεν πρέπει να σταματήσει λόγω αυτών των θεμάτων δυσπιστίας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η επίσκεψή σας είναι πολύ θετική και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να συζητήσουμε σήμερα και αύριο αυτά τα θέματα. Τα συζητήσατε με νομομαθείς, με ειδικούς για θέματα εμπορίου, τώρα και με μας. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε λύση. Θεωρώ ότι το θέμα της προστασίας των δεδομένων θα πρέπει το αργότερο να επιληθεί μέχρι την Άνοιξη. Για να μην έμπλακεί στον τελικό γύρο συζητήσεων για το TTIP, γιατί τότε μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το ήδη δυσχερές θέμα. Και θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων αν μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό και ίσως αν θέλετε κύριε Γερουσιαστά να πάρετε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ και εσά Πρόεδρε Μπροκ και τα μέλη της Επιτροπής σας που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρευρεθούμε σε αυτή τη συνάντηση. Για να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων. Είμαστε μια μοναδική αντιπροσωπεία που ταξιδεύει αυτή τη βδομάδα στην Ευρώπη. Πήγαμε στο Βερολίνο, θα περάσουμε δύο μέρες στη Βρυξέλλη σήμερα και αύριο και θα γυρίσουμε για τη γιορτή των ευχαριστειών στι ΗΠΑ. Είμαστε μοναδικοί γιατί είμαστε μικρή αντιπροσωπεία λόγω των διακοπών, αλλά είμαστε διαπαραταξιακοί και εκπροσωπούμε και τη Γερουσία και το, τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και είμαστε κάποιοι δημοκρατικοί, κάποιοι ρεπουμπλικάνοι και όλοι και οι τρεις μας δηλαδή είχαμε ηγετικέ θέσεις. Εγώ τώρα είμαι πρόεδρος το, της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Ο εκπρόσωπος Μίξ ήταν, είναι δημοκράτης και πρώην ήταν σε αυτήν την επιτροπή στο, στην Βουλή των Αντιπροσώπων και ο άλλος εκπρόσωπος γνωρίζει, γνωρίζεται όπως και είναι πρόεδρος του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου, στο οποίο συμμετέχετε πολύ. Και υποστηρίζουμε φυσικά τις διατλαντικές σχέσεις. Είμαστε ένθερμοι οπαδοί. Θέλαμε να είμαστε σήμερα εδώ σήμερα, ούτω ώστε να ξεκαθαρίσουμε ότι εκπροσωπούμε ε, μια τεράστια ομάδα γερουσιαστών και βουλευτών που θέλουν να κάνουν ό,τι πρέπει, το καταδύναμη, ούτω ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μας ήρθε η ιδέα ε, για αυτό το ταξίδι, γιατί αρχικά ο πρόεδρός σας ε, και κάποια μέλη της Επιτροπής ε, ήρθαν στο Κογκρέσο πριν λίγες εβδομάδες να μας επισκεφτούν και σκεφτήκαμε ότι είναι ευγενικό να κάνουμε και εμείς μία επίσκεψη, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση και συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι μόνο λόγια, αλλά και πράξεις. Πρέπει να υπάρξουν πράξεις. Όπως είπε και ο πρόεδρός σας, η συζήτηση που έχετε τώρα για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και το ρόλο της επιτήρησης ε, στην ε, κοινωνία μας είναι μια συζήτηση που κάνουμε και εμείς στις ΗΠΑ τώρα. Και όντως έχουμε κοινέ ε, αξίες. θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από οποιαδήποτε επιβουλή και οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες ιστορικά ασκούσαν επιτήρηση για να αποτρέψουν διάφορες τέτοιες πράξεις. Ε, το κάνουμε και σε συντονισμό, αλλά ε, συμμεριζόμαστε και την αρχή, την αξία της ε, προστασίας ιδιωτικής σφαίρας. Το να παρισφρίουμε στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών μας δεν μας αρέσει και προσπαθούμε μετά από αυτές τις αποκαλύψεις των πολιτήσεις να παντρέψουμε αυτές τις ανάγκες. Αυτέ οι αποκαλύψει σοκάρισαν του Ευρωπαίου αλλά και του Αμερικανού. Έχουμε ένα σύστημα εποπτεία στο Κογκρέσο ε, των αρχών πληροφοριών, ε, που είναι πολύ αυστηρό, αλλά μόνο λίγα μέλη των ε, λεγόμενων ε, κάποιων κοινοβουλευτικών επιτροπών που λέγονται select committees έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Και μετά από τις αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών κάνουμε στις ΟΠΑ μια συζήτηση για τη χειραγώγηση του μηχανισμού πληροφοριών που κατά την άποψή μας τα τελευταία δέκα χρόνια μεγάλωσε υπερβολικά, έγινε υπερμέγεθες και οι πολίτες μας ζητάνε νέα προστασία, ζητάνε νέες ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε σίγουρα ότι κάποια συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει και νομοθέτημα. Ο Σένσον Μπράνον ε, έκανε μια πρόταση, ο πρόεδρος ε, έκανε μια άλλη πρόταση, αλλά σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω ποια πρόταση θα υπερισχύσει. Ο πρόεδρος είναι πραγματικά α, πολύ, εγκύπτει πολύ σοβαρά στην ανάγκη αλλαγής. Πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι είναι επιφανειακές αυτά, αυτές οι προσπάθειες, αλλά εγώ πιστεύω θα γίνουν και ουσιαστικές αλλαγές. Ε, πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια ε, και για την πολιτική στο Αφγανιστάν και για την στρατιωτική δράση ε, μέσω με εμπιστευτικά, έτσι, όχι προφανή μέσα. Επίσης υπάρχει πρόοδος, πρόοδο, σε διμερείς επαφές μεταξύ μόνο. Και είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την ε, προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και το, την προστασία των εμπορικών συμφερόντων, ε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και θέλουμε να συμμετάσχουμε. Οποιαδήποτε και είναι η πορεία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, θέλαμε πάνω απ' όλα να έρθουμε εδώ σήμερα για να σας πούμε ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτή η σχέση, όχι τώρα μόνο, μακροπρόθεσμα. Και είμαστε δεσμευμένοι να τη βελτιώσουμε. Και νομίζω ότι μόνο μέσω του διαλόγου και ανταλλαγή απόψεων θα βοηθηθούμε ε, και θα βρούμε μια νέα ατραπό. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, να δώσω το λόγο στον Δίας Μπάλαρτ και στον ε, εκπρόσωπο Μίξ για λίγα σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Πρόεδρος της αντιπροσωπείας μας. Ένα ωστόσο σημείο θέλω να το επαναλάβω, το γεγονός ότι είμαστε τόσο δεσμευμένοι στη σχέση αυτή. Δεν χρειάζεται να σας πω. Εδώ, σε εσά τους βουλευτές. Ότι η δημοκρατία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και ότι οι δημοκρατίες είναι ατελείς μη τέλειες. Η σχέση μας δεν είναι η πρώτη φορά που υπόκειται πίεση, ούτε θα είναι η τελευταία άλλωστε που υπόκειται πίεση. Γνωρίζουμε όμως, όπως και εσείς ε, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, ότι η καλύτερη εγγύηση, η εγγύηση ελευθερίας, η εγγύηση ασφάλειας, η εγγύηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κρατούς δικαίου, είναι ακριβώς η δύναμη της σχέσης αυτής της διατλαντικής σχέσης. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όπως είπε και η η συζήτηση και οι ανησυχίες που εκφράζονται εδώ από τους φίλους μας στην Ευρώπη είναι ακριβώς οι ίδιες που αντιμετωπίζουμε και συζητάμε στην Αμερική, στο Κογκρέσο. Και παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία είναι ατελής, είμαι και εγώ πεπισμένος ότι και πάλι ο Πρόεδρος κάνει μια πολύ σημαντική αναθεώρηση και ας είμαστε ειλικρινείς. Αν η αναθεώρηση αυτή δεν αποδώσει με σοβαρό τρόπο και με πεπισμένο ότι πρόκειται να αποδώσει, ο Πρόεδρος θα υποστεί πολλές πιέσεις από... και από τις δύο, και από το... την Γερουσία και από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό καταδεικνύει ότι το παίρνουμε αυτό στα σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερο στην κυβέρνηση, το παίρνει στο, πολύ στα σοβαρά το Κογκρέσιο, αλλά και πάλι ο σκόπο τη επίσκεψή μα είναι να εκφράσουμε εκ νέου τη σημασία που έχει για μα αυτή η σχέση. Αποτελεί την καλύτερη, την πιο ακλόνητη εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ασφάλεια, για το κράτο δικαίου. Αυτό προκύπτει από τη διαρκή προσπάθεια ενδυνάμωση της σχέση αυτής. Πρόκειται για ένα προνόμιο και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να περάσουμε λίγο χρόνο εδώ στην Επιτροπή σας με ομόλογους μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο, κύριο Μίξ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με το μήνυμα αυτό που απέφτυναν οι προλύσαντε. Εμεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, στο Κογκρέσο αλλά και ο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών κατανοούμε τη σημασία τη σχέση αυτή. Επίση κατανοούμε την αξία τη εμπιστοσύνη και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό που συνέβη για να ανεκοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη ένθεν και του Ατλαντικού. Μια εμπιστοσύνη που εδώ και καιρό χαρακτηρίζει τις σχέσεις των χωρών μας, των μεγάλων μας χωρών. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό για μας που είμαστε εδώ σήμερα, για να, σας, ε, για να μεταβιβάσουμε στην Αμερική τα μηνύματα που θα μας δώσετε, αλλά και για να σας μεταβιβάσουμε το δικό μας μήνυμα, ότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε το λαό μας ασφαλή, ούτε να έχουμε μια δημοκρατία χωρίς τη δική σας βοήθεια. Ο κόσμος έχει αλλάξει και μόνο από κοινού θα καταφέρουμε να τα διορθώσουμε αυτά. Σε μια εποχή νέας τεχνολογίας, κοινωνικών μέσων, κοινωνικών μίδια, μια εποχή του διαδικτύου, πρέπει από κοινού να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν μπορούν οι ΙΠΑ να τα κάνουν μόνοι τους αυτά. Ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες να τα κάνουν μόνοι τους. Από κοινού θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε σε κάθε περίπτωση να σας μεταβιβάσουμε, ότι για μας έχει σημασία αυτή η σχέση. Είναι σημαντική για μας. Και αυτό που συνέβη και προκάλεσε αυτή τη ρήξη στην εμπιστοσύνη είναι κάτι που ο λαός της Αμερικής το παίρνει πολύ στα σοβαρά. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να σπρώξουμε κάτω από το χαλί. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση και ως λαός. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό που έχουμε από κοινού είναι οι αξίες. Οι αξίες της δημοκρατίας, οι αξίες ε, της διασφάλισης των ελευθεριών, η αξία της ιδιωτικής σφαίρας, η αξία της ε, ασφάλειας των πολιτών. Χαιρόμαστε λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας και για να ε, βεβαιωθούμε ότι θα παραμείνει αυτός ο ισχυρός δεσμός που έχουμε και μάλιστα για πάντα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Αλαφρανκά. Ευχαριστώ. Από πλευρά της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, γερουσιαστή Μάρφη και του αντιπροσώπου Δίαθ Μπαλάρ και Μίξ που είναι ε, καλή φίλη πολλών ε, μέλων του Κοινοβουλίου εδώ και πολλά, του Κοινοβουλίου εδώ και πολλά χρόνια. Και την ε, ε, επίσκεψή σας θεωρούμε δείγμα επίδειξης και ενδιαφέροντος για την, τις σχέσεις με την Ευρώπη. Θα είμαι πολύ σύντομος μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε και σήμερα στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών της ειδική Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, πολλοί πιστεύουμε ότι η διατλαντική σχέση είναι στο γονιδίωμα της Ένωσης. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, αυτή η σχέση έχει τρωθεί. Ξέρετε ότι αυτά τα θέματα κατασκοπίας οδήγησαν ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου να ζητήσουν να ε, ανασταλεί η συμφωνία SWIFT και ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να ανασταλεί και η συμφωνία Βένερ. Άρα χρειάζεται μια καθαρή, σαφής απάντηση για να επανέλθουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Όπως ακούσατε, σήμερα το πρωί η Αντιπρόεδρος ε, Ρέντινγκ προετοιμάζει μια πολιτική δήλωση και η επίσκεψή σας γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σκόπιμη. Αυτό που θέλουμε λοιπόν από εσά είναι συγκεκριμένες απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ούτως ώστε στη βάση αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και διαλόγου να διορθώσουμε την κατάσταση και να ε, ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους τον ε, γερουσιαστή και τα δύο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους για μας. Οι αποκαλύψεις του πρώην κατασκόπου Σνόντεν καταράκωσαν πλήρως την εμπιστοσύνη προς ε, την ε, κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και προς τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Αλλά δεν ήταν το πρώτο γεγονός αυτό που ε, έφυξε αυτήν την εμπιστοσύνη. Και προηγουμένως είχαμε κάποια δείγματα για προβλήματα εμπιστοσύνη σε σχέση με τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει Σουίθ και Βενεργέτη. Στην πρόσφατη επίσκεψή μας η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών την επίσκεψη που κάναμε λοιπόν το Μάρτιο 2012 δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε δυστυχώς με τα μέλη του Κογκρέσου και σημειώσαμε ότι η θέση τους ήταν μια θέση έλλειψης κατανόησης για το τι σημαίνουν τα ευρωπαϊκά μας συντάγματα και η αξία, η σημασία που αποδίδουμε στον ε, ιδιωτικό βίο, στην ιδιωτική σφαίρα. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε διαφορετικές παραδόσεις, αλλά βεβαίως Πρέπει να καταπολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Είμαι Ισπανίδα. Έχουμε υποφέρει πολλά από την τρομοκρατία. Αλλά πάντα προσέξαμε η καταπολέμησή της να γίνει πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας. Για μας η πρόληψη της ε, τρομοκρατίας και γενικά της εγκληματικότητα δεν μπορεί να γίνεται με βάση την αρχή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η μαζική συλλογή στοιχείων χωρίς καμία δικαστική έγκριση, τουλάχιστον με βάση τη δική μας αντίληψη για το Σύνταγμα και τη δικαστική ένωμη τάξη. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι αστυνομικού τύπου αν γίνεται κάτι τέτοιο. Και αυτό όχι μόνο ε, εισέρχεται στα δικά μας θέματα ιδιωτικού βίου, είναι μια κυβέρνηση η οποία ε, και στο εμπορικό μας σύστημα ανταλλαγών ε, μπορεί να παρεμβαίνει και παρεμβαίνει και στην ε, πολιτική μας διαδικασία διαμόρφωση απόψεων. Ελπίζω να μπορέσει να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Σας προτείνω 1,5 λεπτό κάθε ομιλητή, γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Τώρα, η Βαρόνι Λάτφεντ, που ελπίζω να δώσει καλό παράδειγμα τήρηση του χρόνου. Ναι, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Βασίλη Τσουέρτ και τα δύο μέλη τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Δία Μπαλάρτ και Μίξ, ξέρουμε. Πολύ εξημών, πολύ καλά τον Δία Μπαλάρτ, που ήταν αντιπρόεδρο τη Αντιπροσωπεία ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε συνεργαστεί μαζί του και συμμετέχω ε, στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και Δικαιοσύνη για θέματα προστασία ε, δεδομένων και νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση ενώπιον μας και είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ και που αντιμετωπίσετε σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε μία νέα γενική συμφωνία. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές πλευρές, ε, το εμπόριο, προστασία δεδομένων, θέματα συλλογής προφοριών και ε, ε, υπάρχουν και θέματα αρμοδιοτήτων εδώ. Αλλά εάν δεν λύσουμε το θέμα μαζί, θα καταρρεύσουμε ο καθένας και χωρισμένα. Υπάρχουν διάφοροι εδώ στις Βρυξέλλες που με κάπως ανεύθυνο τρόπο καλούν να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις TTIP. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να κρατάμε τα δεδομένα μας εντός της Ευρώπης. Θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος. Δεν θα τα ε, μεταφέρουμε. Αυτό βέβαια είναι στην ουσία κάπως προστα... αντίληψη προστατευτισμού. Βέβαια αυτή δεν είναι η κατεύθυνση που θέλει η ομάδα μου να ακολουθηθεί. Αλλά από αυτή την κρίση πρέπει να βρούμε μια δυνατότητα να καταλήξουμε σε κάποια θέματα που εδώ και καιρό μας απασχολούν. Για το πώς δηλαδή θα έχουμε το σωστό πλαίσιο εμπιστευτικότητας και από πλευράς νομική και από πλευράς εμπορικών συμφερόντων. Οπότε επαναλαμβάνω το μήνυμα που εσείς μας αποστέλλετε. Θα έπρεπε να γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσει μια σωστή συζήτηση και στο Λονδίνο θα τα σκόπω, συζήτηση που γίνεται και διακόπτει ο Πρόεδρος. Δυστυχώς δεν, ακούμε το, δεν υπάρχει μικρόφωνο ανοιχτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε Χίρς. Εγώ είμαι από τη Γερμανία και είμαι και μέλος της αντιπροσωπείας με τις ΗΠΑ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ήρθατε εδώ σήμερα και ιδιαίτερος επειδή ήσασταν και χθε στο Βερολίνο και ήταν μεγάλο το θέμα αυτό που συζητήθηκε. Ε, ήταν πραγματικά έντονη η εκτίμηση και χαίρομαι και που βρίσκατε και στις ε, Βρυξέλλες. Το θέμα λοιπόν ε, είναι ότι είναι σημαντική η σχέση μεταξύ Βερολίνου και ΕΙΠΑ. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι στην Γερμανία ιδιαίτερως είναι μεγάλη η αγανάκτηση με αυτά που μάθαμε τους τελευταίους μήνες και αναστάτως. Είναι καλή ένδειξη, θεωρώ, το γεγονός ότι θέλετε να γίνει διάλογος και συζητώ και με πολλούς ε, νέους και στο facebook και στο ίντερνετ και αναφέρουν τις αμφιβολίες τους γιατί λένε για παράδειγμα ότι α, όταν πηγαίνουμε στη ΣΥΠΑ αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά εδώ μας άρα θα πρέπει να προειδοποιηθούμε ότι θα πρέπει να οικοτομήσουμε εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ όπως και η συνάδελφος είπε πριν από λίγο, θεωρώ ότι με τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου πάμε σε ένα καλό δρόμο, οδεύουμε προς μια καλή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσει να είναι ένα σημαντικό τμήμα αυτό η προστασία των δεδομένων της ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Από την ομάδα του ECR είμαστε η πιο μεγάλη ομάδα σε ό,τι διαφορά αυτό το θέμα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα σχέση με τη ΣΥΠΑ. Ο Καναδάς, Εθνική Αμερική, Μεξικό, Κολομβία, Χιλή και η Βραζιλία από την άλλη πλευρά. Θεωρούμε ότι εκεί το μέλλον είναι ό,τι αφορά αυτή την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, το TTIP σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το ελεύθερο εμπόριο από τη δική σας πλευρά του Ατλαντικού και πέρα από τον Ειρηνικό. Και ανησυχούμε με τις, αυτά που ακούγονται για να σταλούν οι συζητήσεις για το TTIP. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς κοινού συμφέροντος. Εγώ έρχομαι από το Μαυροβούνιο γιατί είμαι συγκεκριτή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουν να προσκληθούν στο ΝΑΤΟ περιμένουν αμερικανική πρόσκληση. Άρα υπάρχει μια κοινή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με την επιρροή λοιπόν από την κυβέρνησή σας. Σας παρακαλώ κάντε κάτι και για το Μαυροβούνιο. Πρόκειται για μια δημοκρατία που έχει τις ειδικέ μας αρχές και αξίες και είναι και υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο ειρήνευση τη Μέση Ανατολή, τα κουαρτέτο Γενεβαδίο για το Ιράν, ε, Βορειά Κορέα, Κίνα, Κινέζικη θάλασσα, Συρία, όλοι αυτοί είναι τομεί όπου χωρί την Αμερικανική συνεργασία, χωρί μια κοινή ηχηρή φωνή, ιδιαίτερα στη Συμβούλια Ασφαλεία, δεν θα πάνε πολύ μακριά τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την NSA. Σχόλιο εκτό μικροφώνου του Προέδρου. Να, πω, να κάνω μία παρατήρηση, να πούμε ίση αντιμετώπιση των Ευρωπαίων ε, υπηκών στα δικαστήρια τα Αμερικανικά. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά μέσα, σε ό,τι αφορά. Κύριε Σταγκουράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για τους επισκέπτε από τις ΗΠΑ... οφείλω να του πω ότι αντιπροσωπεύω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έρχομαι από την Ελλάδα, και θα ήθελα να του πω το εξή. Ε, καταρχήν, νομίζω ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα συμφωνούμε ότι αυτό που έγινε έγινε με πολιτική απόφαση. Υπήρχαν συγκεκριμένες πολιτικές που οδηγήσαν συγκεκριμένα, στα συγκεκριμένα μέτρα. Το θέμα δεν αφορά μόνο την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Το θέμα αφορά έναν πόλεμο θα έλεγα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους σε πολλά πεδία και στο πεδίο των πληροφοριών, όπως μάθαμε από τον τύπο. Δεύτερον, ε, χάρη στις αποκαλύψεις του Σνόντεν, και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Είπατε ότι έχει σοκαριστεί η αμερικάνικη κοινή γνώμη για την κατασκοπία που γινόταν. Αλλά δεν βλέπω η αμερικάνικη, η αμερικάνικη κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον Σνόντεν με θετικό τρόπο. Αντίθετα, πολλοί στη χώρα σα τον θεωρούν προδότη. Εν πάση περιπτώσει, χάρη στι αποκαλύψεις αυτές μάθαμε ότι παρόμοιε πρακτικέ ακολουθούν και πολλέ υπηρεσίε των ευρωπαϊκών χωρών. Άρα το αμάρτημα δεν είναι μόνο των ΗΠΑ, είναι και των ε, κυβερνήσεων των χωρών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα είναι φανερό γιατί γίνεται αυτό, γιατί και οι δύο είναι ε, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουμε καπιταλιστικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν σέβονται τελικά ούτε ανθρώπινα δικαιώματα ούτε ελευθερίες όπως αποδείχθηκε τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Τρίτον, θα ήθελα να ασκήσετε την επιρροή σας για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Το πρώτο είναι η άρση του εμπάργου κατά της Κούβας, ένα άδικο εμπάργο και δεύτερο την επιρροή σας στην απελευθέρωση των πέντε Κουβανών οι οποίοι, οι οποίοι αδίκως κρατούνται όπως ξέρετε στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών. Danke, ε, Herr Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, τους Αμερικανούς φίλους και τονίζω το αυτό το φίλους να ξέρουν πόσο σκεφτόμαστε εμείς ε, οι χριστιανοδημοκράτες. Είμαι εδώ και 35 χρόνια στο Κοινοβούλιο και ήμουν επί σειρά ετών επικεφαλής της ομάδας μου και ε, πλήττομαι πραγματικά από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι μυστικέ υπηρεσίε τη Αμερική. Είσαστε ένα κράτο δικαίου και σε ένα κράτο δικαίου δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ένα δεύτερο θέμα ήθελα να αναφέρω. Γκουαντάναμο. μου. Τόσα χρόνια καταπιέζεται. Είμαι υπέρ τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Δεν μπορεί όμω κανεί να φυλακίζει επί σειρά ετών χωρί ε, προσαγωγή άτομα, χωρί να έχει αποδείξει, χωρί να του έχει δικάσει ότι είναι τρομοκράτε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ κατεπηγόντως να επιλύσετε τα θέματα αυτά και να κάνετε τα απαραίτητα για να ελέγξετε τις μυστικές σας υπηρεσίες. Και αυτό το περιμένουμε από εσά γιατί είσαστε φίλοι μας, γιατί αν καταρρεύσει το κράτος δικαίου θα καταρρεύσει και η δημοκρατία τελικά. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο συνάδελφος από τη Νέα Υόρκη, ότι αυτή η σχέση μετράει. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε από εσά, γιατί από άλλου μπορεί να τα περιμέναμε αυτά, όχι όμω από τι ΗΠΑ. Ο κ. Σαρλάκη. Ευχαριστώ, γερουσιαστή Μέρφυ. Εκτιμώ τα όσα είπατε. Και αυτό που είπατε αρχικά για το τι χρειάζεται να γίνει για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Να σας δώσουμε απλές απαντήσεις από ευρωπαϊκής πλευράς. Καταρχάς, διαλύστε αυτόν τον τεράστιο μηχανισμό επιτήρησης που έχετε. Δεν είναι δημοκρατικό, δεν προστατεύει αλλά καταστρέφει τις πολιτικές ελευθερίες και δεν χρησιμεύει για να καταπολεμήσει τη τρομοκρατία. Δεύτερον, να μάθετε από την ευρωπαϊκή εμπειρία ε, και τον τρόπο που καταπολεμούμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Είχαμε τρομακρατικό πρόβλημα στην δεκαετία του 80 στην Ήπειρό μας, πολύ μεγαλύτερο το δικό σας και το αντιμετωπίσαμε χωρίς να χτίσουμε αυτούς τους τεράστιους μηχανισμούς, χωρίς να περιστύλουμε τις αστικές ελευθερίες, χωρίς να βάλουμε τέτοιες ε, συνοπτικές διαδικασίες δίκης, τέτοιες ποινές και καταφέραμε να μην είναι μείζωνα ε, απειλή η απειλή της δημοκρατίας σήμερα. Στην Ιταλία και σε άλλες χώρες παλέψαμε την δημοκρατία με τα εργαλεία που μας δίνει η δημοκρατία. Με δίκαιες δίκες. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί. Σε μία Ήπειρο που πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερη στις ΗΠΑ. Μάθατε λοιπόν από τη δική μας εμπειρία. Ούτως ώστε να είμαστε και φίλοι στο μέλλον. Αν το κάνετε θα παραμείνουμε φίλοι. Mr. Ευχαριστώ τους διακεκριμένους επισκέπτες μας. Σας ευχαριστώ και για την ε, φιλοξενία σας στην Ουάσιγκτον. Ε, Θέλουμε να τα ανταποδώσουμε τρεις εβδομάδες μετά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό ε, έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών, όχι μόνο στις ΗΠΑ και στις χώρες μας. Είναι κοινή πρόκληση αυτή και πρέπει να κάνουμε και δύο τη δουλειά μας. Και είναι πρόβλημα και για τα εθνικά κοινοβούλια στις χώρες μας. Θέλω να πω τώρα κάτι για το μέλλον. Η συμφωνία TTIP είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά φοβάμαι ότι οι λαοί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν συνειδητοποιούν τη σημασία αυτής της συμφωνίας και ότι στο μέλλον, χάρη σε αυτή τη συμφωνία, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας, θα επεκταθεί η οικονομία μας και ελπίζω να μπορέσετε να στείλετε αυτό το μήνυμα και στους Αμερικανούς όταν επιστρέψετε. Ο κ. Στάνοκ ανέφερε κάτι για την σταθερότητα στην Ευρώπη που είναι πολύ σημαντική και ανέφερα και το Μαυροβούνιο. Το είχαμε πει και στη Ουάσιγκτον όταν είχαμε έρθει. Η διεύρυνση θα φέρει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, Λαμβάνοντα τι αρνητικέ εξελίξει στην Ουκρανία υπόψη, ε, πρέπει να δώσετε μια ευκαιρία ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Thank you for coming to the Ευχαριστώ που ήρθατε στο Κοινοβούλιο συμφωνούμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί, γιατί αυτή η σχέση έχει σημασία και γιατί έχουμε τις ίδιες αξίες. Το θέμα είναι, έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Ε, στην πρόσφατη επίσκεψή μας στην Ουάσιγκτον μάθαμε ότι οι Αμερικανοί δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, ενώ οι Ευρωπαίοι στην ιδιωτική σφαίρα. Επίσης, ε, κάποιοι Αμερικανοί ε, αμφισβητούν έννοιες όπως η ιδιωτική σφαίρα. Αυτές διαφορές, πώς τις βλέπετε, υπάρχει βάση για να καταλάβουμε οι μεν τους δε. Δεύτερον, έχετε αυτό αυτή την νομοθετική πράξη, το ΦΑΙΣΑ. Ε, ε, με τους γείτονές σας έχετε συμφωνήσει να μην κατασκοπεύετε οι μεν τους δε. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό και με τους Ευρωπαίους φίλους σας και συμμάχους σας. Σας ευχαριστώ και καλωσορίζω τους φίλους μας. Δεν θέλω να αλλάξω το θέμα. Συγγνώμη, θέλω να αλλάξω το θέμα. Πότε θα αντιμετωπίσετε τις, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ με τον ίδιο τρόπο. Μιλάω για τη Μέση Ανατολή. Έχετε πάει ποτέ κάποιος από εσά στην Παλαιστίνη για να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Ένα τελείως διαφορετικό θέμα ήταν αυτό. Danke, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ κύριε Σπίρκερ. Οι συζητήσεις που διεξήγαμε, οι συζητήσεις που κάναμε στην Ουάσιγκτον θεωρώ ότι ήταν και επικοτομητικές και ανοιχτού χαρακτήρα. Σας ρωτώ λοιπόν, μάλλον δεχτήκατε την πρόσκληση και το γεγονός ότι υπάρχουν τακτικές επαφές μεταξύ ημών θεωρώ ότι είναι καλό για να αποφευχθούν οι πιέσεις και οι τριβές. Είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την πρόληψη, είναι πάρα πολύ σημαντική και θετική. Έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν αυτές οι ενοχλήσεις ε, λόγω της ε, NSA και αναφέρθηκε ότι όταν ε, ήμασταν στις ΙΠΑ υπήρχε η αίσθηση ότι αγνοείται, ότι δεν τηρούνται οι, δεν νόμοι και ότι είμαστε εκτός ελέγχου. Διαρκώς ρωτώ λοιπόν πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το Freedom Act και για να ανοικοδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, να αποκαταστήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, πώς μπορούμε να βρούμε λοιπόν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία των ε, υπηρεσιών αυτών, προκειμένου να ξαναρχίσουμε αυτή τη συνεργασία βάσει εμπιστοσύνης με τη ΣΥΠΑ. χωρίς όμως ε, τις ενοχλήσεις αυτές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες εκδηλώθηκαν. Thank you, Mr. Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γερουσιαστά, κύριε. Είμαστε, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σημαντικός αυτός ο διάλογος. Σας καλωσορίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε την ευθύνη να μιλήσουμε για τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να γίνουν από εμάς τους νομοθέτες και να σκεφτούμε. Καλό θα ήταν, πέρα από αυτά τα οποία αναφέρετε, πείτε μας ε, τι κάνετε και στη Γερουσία και στο Κογκρέσο για να ξεπεράσετε αυτή, αυτές τις υπερβολές από πλευράς της NSA. Θεωρώ ότι είναι δική μας ευθύνη να σκεφτούμε το τι γίνεται προκειμένου να περιορίσουμε τις αυτερεσίες κάποιων μυστικών υπηρεσιών. Κοιτάξτε, εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου στην Ανατολική Γερμανία είχαμε παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν. Μου δημιουργεί λοιπόν ένα περίεργο ντεζαβού αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτές τις δημοκρατίες, σε ό,τι αφορά την υπηρεσίες αυτές. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι της ιστορίας, αυτό το κομμάτι του παρόντος θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλαμ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας, για τη συνεργασία σας. Η ασφάλεια αποτελεί μια κοινή πρόκληση στον σύγχρονο κόσμο είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας μόνος του. Και ε, βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Τι γίνεται όμως όταν έχει ε, τρωθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Αυτό που με ανησυχεί είναι η άνηση μεταχείριση σε ό,τι αφορά την παροχή αγγίσεων, ε, σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε μια ισόρροπη προσέγγιση. Η παρουσία σας εδώ αποτελεί μια εγγύηση ότι μπορούμε εκ νέου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουν. Είναι ιστορική η ευθύνη που φέρουμε και είμαστε και οι δύο πλευρές υπεύθυνε επιφορτισμένες και συμφωνώ ότι το SWIFT δεν θα πρέπει να ανασταλεί. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ που ήρθατε. Είδα όταν ήμουν πριν από τρεις εβδομάδες στη Washington, είδα πόσο πιστεύουν στις αρχές της Διατλαντική Συμφωνίας οι συνομιλητέ μας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση και να σας κάνω ένα σχόλιο. Ερώτηση. Πότε θεωρείτε ότι η διαδικασία αναθεώρηση που ζήτησε ο πρόεδρος Ομπάμα θα καταλήξει και προς τα που πάει. Και σχόλιο. Μια διατλαντική σχέση τόσο σημαντική πρέπει ακριβώς να συνοδεύεται και από θετικά σύμβολα. Για παράδειγμα η ετήσια συνάντηση κορυφής είναι πολύ σημαντική. Και τώρα που έχουμε και έναν μόνιμο πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Φανρόμπουη, που ήταν για πέντε χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ήδη από την εποχή του Προέδρου Κλίντον είχαμε αυτές τις συναντήσεις, αλλά στην πράξη δεν, γίνονται τώρα με τον ε, πρόεδρο Ομπάμα. Θα πρέπει να καταλάβει η Ουάσιγκτον ότι πρέπει να έχουμε θετικέ εικόνε. Όπω για παράδειγμα μέσα τη κορυφή. Αυτό το μήνυμα να μεταφέρετε, παρακαλώ. Ο κύριος Μάρφιν, Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τις ανησυχίες σας, ε, τα αισθήματα. Πολύ σύντομα θέλω να απαντήσω μερικά από τα θέματα που θίξατε. Και θα αφήσω του συναδέλφους μου να απαντήσουν σε ορισμένα άλλα. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι κυρίως συζητάμε για δύο διαφορετικά και αρκετά απομακρυσμένα θέματα. Το ένα είναι θέμα πολιτικής ε, κατασκοπίας, δεν θέλω να μιλήσω για τους ε, εκ μέρους των άλλων, αλλά νομίζω ότι πολλοί στο Κογκρέσο θεωρούμε ότι όντως παραβιάσαμε ορισμένες αρχές. Πήγαμε στη Γερμανία πριν έρθουμε εδώ, συγκεκριμένα γιατί ξέρουμε το θέμα ότι έχει θυγεί η εμπιστοσύνη λόγω των παρακολουθήσεων του τηλεφώνου της Καγκελαρίου. Και ελπίζω ένα από, ένα από τα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης που την περιμένουμε πριν το τέλος του χρόνου να είναι ουσιώδης αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε την πολιτική μας επιτήρηση. Βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι που κάνουμε τέτοια επιχειρήση, αλλά είναι σαφές ότι η σχέση ωφέλους ε, ε, και κόστους ε, δεν ήταν αυτή που αναμέναμε. Θα θέλαμε λοιπόν να χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές. γιατί ξέρουμε ότι συλλέγησαν στοιχεία, σε μεγάλο βαθμό σε συντονισμό με τις δικές σας υπηρεσίες πληροφοριών, με τα δεδομένα. Αυτό καλύτερα να γίνεται σε διμερή βάση. Γιατί στο βαθμό που εφήγει η ιδιωτική σφαίρα, η λύση είναι να υπάρχουν καλύτερες διαδικασίες και από πλευράς των Αμερικανικών υπηρεσιών ε, πληροφοριών, αλλά και από την πλευρά των ε, υπηρεσιών των ε, κρατών της Ένωσης. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Διμερός βεβαίως. Δεύτερον, Εκτιμώ τα σχόλια όσων είπαν ότι δεν θα έπρεπε να συσχετίσουμε υπάρχουσε συμφωνίες που ε, μας βοηθάνε στην προστασία, για παράδειγμα, η βάση δεδομένων για τα στοιχεία των επιβατών, των πτήσεων και του SWIFT και επίσης αυτούς που είπαν ότι δεν πρέπει να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις για το TTIP. Ήρθαμε για να καταστεί σαφές ότι δεν χρειάζεται να αποστείλετε και περαιτέρω μήνυμα θέτοντας σε κινδύνο την συλλογική μας ασφάλεια μέσω της αναστολής αυτών των συμφωνιών. Εμείς πιστεύω ότι το Κογκρέσο ειλικρινά προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να υπερβούμε το πρόβλημα ενώ εφαρμόζουμε και διαπραγματευόμαστε συμφωνίες. Τρίτον, όλοι είμαστε το προϊόν της συλλογικής μας εμπειρίας. Ε, βεβαίως ε, έχουν υπάρξει τρομερές τρομοκρατικές ενέργειες. Ε, δεν θα συμφωνώ ότι είναι απειλή στην Ευρώπη η τρομοκρατία σήμερα. Ακόμη αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις ε, από τη δολοφονία χιλιάδων Αμερικανών από τη μεγαλύτερη τρομοκρατική απόπειρα που έγινε ποτέ στο έδαφο μα και αυτό ήταν και αποτυχία των μυστικών μα υπηρεσιών. Αυτό που συνέβη έκτοτε είναι μια τρομερή εξάπλωση των μυστικών μα υπηρεσιών. Τώρα λοιπόν πρέπει να βρούμε ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθό του. Αλλά αυτό που έγινε πριν από πάνω από μια δεκαετία είναι η βάση τη ε, έκτοτε εξέλιξη. Και τώρα λοιπόν πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό που κάναμε έκτοτε γιατί η πείρα μας είναι φυσικά, το παρελθόν μας είναι και η προστασία των δημοσίων ελευθεριών. Κάνουμε λοιπόν σοβαρές συζητήσεις. Έχουν να κάνουν με νέους νόμους που θα επέτρεπαν ε, οι πληροφορίες που παίρνουν τις δικαστικές εντολές για να αποστέλουν στοιχεία να μπορούν να τις κοινοποιήσουν. Υπάρχουν επίσης και οι προτάσεις του γερουσιαστή Λύχη που στην ουσία θα απαγόρευαν την συλλογή μεταδεδομένων. Υπάρχουν όμως πολλοί στις ε, αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που θεωρούν ότι πάνω από 50 τρομοκρατικές απόπειρες αποφέρθηκαν λόγω της συλλογής αυτών των στοιχείων. Τελευταίο. Ο καθένας προσπαθεί και αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις ε, απειλές κατά της χώρας του. Μπορούμε να προσπαθούμε να καταδιώξουμε παντού τους τρομοκράτες και να κάνουμε τεράστιες ε, προσπάθειες συλλογής στοιχείων για να τους πιάσουμε, να τους βρούμε και να τους πιάσουμε. Αλλά επιπλέον μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους λόγους για τους οποίους μπορούν να στρατολογούν οι τρομοκράτες για τις ε, απόπειρές τους. Και τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε και εμείς και οι σύμμαχοί μας αυτό που θα κάνουμε λοιπόν και εμείς και οι σύμμαχοί μας για να σεβαστούμε τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα προστατεύσουμε τις χώρες μας. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ προστασίας ε, της ασφάλειας της χώρας μας και προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών. Δεν επαρκεί η συλλογή στοιχείων και η επιτήρηση. Πρέπει να μειωθούν, να μειωθούν οι λόγοι για του οποίου διάφοροι είναι εναντίον μας και προσπαθούν να οργανώσουν επιθέσεις εναντίον μας στον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα. Υπάρχει μία ομάδα στο Κογκρέσο που ειλικρινά πιστεύει πως αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθηθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απαντήσω κι εγώ για τις διαφορές στη συμπεριφορά μας και για το πώς βλέπετε εσείς και εμείς την ασφάλεια και την ιδιωτική σφαίρα όλοι προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Ε, η ιδιωτική σφαίρα χωρίς ασφάλεια δεν σε οδηγεί πουθενά. Ενώ ασφάλεια χωρίς ιδιωτική σφαίρα επίσης δεν σε οδηγεί πουθενά. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε αυτή τη λεπτή ισορροπία. Και βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη την εμπειρία μα ο καθένα και την πραγματικότητα με στην οποία ζούμε ο καθένα. Η μνήμη τη 11η ε, ε, Σεπτεμβρίου είναι νοπίστη ακόμα. Έχουμε υποφέρει τρομερά από τρομοκρατικέ απειλέ και εμεί, αλλά ξέρω ότι και η Ευρώπη έχει υποφέρει τρομερά από τρομοκρατικέ απειλέ. Και η επίθεση στη Βοστόνη επίση είναι πολύ φρέσκια στη μνήμη μα. Όπω είπε και ο πρόεδρο τη προσωπία μα, υπάρχει το θέμα του TTIP και του SWIFT. Το αναφέρατε πολύ από εσά. Είναι δύο θέματα πολύ σημαντικά για τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά είναι πολύ σημαντικά και για την Ευρώπη. Το ίδιο σημαντικά και το τονίζω, το υπογραμμίζω, ίσως και πιο σημαντικά. Αν πιστεύετε στην ελευθερία και στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο, στο κράτος δικαίου, αυτά θα αλλάξουν τον κόσμο. Να μην ξεχνάμε λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο. η εμπιστοσύνη. Το ακούσαμε, το ξανακούσαμε, φυσικά έχει τρωθεί. Και ένα από τα σημαντικά πράγματα που θα το πούμε και θα το ξαναπούμε εμείς οι Αμερικανοί είναι ότι είμαστε εδώ σήμερα γιατί ξέρουμε ότι έχει συμβεί αυτό. Ε, για να ξαναποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και να τους συμπεριφερόμαστε φιλικά. Και να ξέρουμε βεβαίως και ποιοι είναι οι εχθροί μας και να τους αντιμετωπίζουμε ως τέτοιους. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Σε αυτό που είπε ο κύριος Μιλάν Μον και στην πρόταση που έκανε μιας συνόδου κορυφής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, πολύ συγκεκριμένη, την οποία θα διαβιβάσω στους Αμερικανούς ομολόγους μου. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ιδέα. Ακούστηκαν πάρα πολλά σχόλια. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω. Εν θα ήθελα να πω το εξή. Θέλω να επανέλθω εκεί που, από που ξεκίνησα. Η δημοκρατία είναι ατελής. Στην δημοκρατία απλώς μπορούμε να διορθώσουμε τις ατέλειες, χωρίς να φοβόμαστε τα αντίπεινα και την τιμωρία. Κάποιοι μίλησαν για καπιταλιστικές χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα. Αλλά θέλει κανένας να ανταλλάξει τις ατέλειες της δημοκρατίας και την ελευθερία αυτή με την ουτοπική με την τοπία της κομμουνιστικής Κίνας ή του κομμουνιστικού Βιετνάμ ή της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας. Ξέρω ότι η απάντησή σας είναι όχι. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την φιλία σας. Σας ευχαριστώ που μας δεχτήκατε εδώ στην Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ντις ανέφερε αυτά που θέλω να πω και εγώ για τη δημοκρατία. Κοιτάξτε, είναι μία από τις πιο άτακτες μορφές διακυβέρνησης που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, αλλά αποτελεί την καλύτερη μορφή διακυβέρνησης την οποία εγώ γνωρίζω και ακούγοντας τους ομιλητές σήμερα, βλέπω τη δημοκρατία πώς λειτουργεί στην πράξη. Ακούω διαφορά και διάσταση απόψεων. Σε μία επιτροπή όπου είσαστε ελεύθεροι να μιλήσετε για τις διαφορετικές σας απόψεις και γίνεται συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής όταν δεν είμαστε εδώ που φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ έντονες και θερμές διαστάσεις και διαφορετικές απόψεις. Και γιατί το αναφέρω αυτό. Για να απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις σας. Πότε θα σταματήσουν αυτές οι... Πότε θα κάνει κάτι το κογκρέσο. Θέλω να ξέρετε ότι ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει διαφορά απόψεων και για να καταλήξουμε σε μία συνένεση θα πάρει χρόνο. Έχουμε διάφορα νομοσχέδια. Γιατί ο κόσμος έχει πληχθεί και έχει ισοκαριστεί από το θέμα της NSA στην Αμερική, αλλά υπάρχουν διάφορες σκέψεις για το πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε και να αντιδράσουμε. Και στη ΣΥΠΑ θέλω να ξέρετε σήμερα δεν βασιζόμαστε σε τέτοιες απόψεις βάσει του κόμματός μας, του πολιτικού μας κόμματος. Οι, τα νομοσχέδια που συζητιούνται δεν βρίσκουν σύμφωνα τα κόμματα. Κάποιοι από τους πιο συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους, κάποιοι από τους φιλελεύθεροι, υποστηρίζουν το ίδιο νομοσχέδιο. Και ύστερα κάποιοι άλλοι, στη μέση, τώρα δεν ξέρω προς τα πού να στραφούν. Ποιους να υποστηρίξουν. Σας είπα Ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις κάποια πράγματα τα υποστήριζα σε μια προεκλογική εκστρατεία και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το... δεν τα υποστήριζα. Το Patriot Act, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει η δημοκρατία. Μαθαίνω από τις εμπειρίες μου για το τι πρέπει να κάνω, τι είναι το σωστό να κάνω. Και αυτή λοιπόν είναι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον και στην Αμερική. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερω είναι το εξή. Δεν θέλω να θεωρήσετε το γεγονό ότι γίνεται καν αυτή η συζήτηση στην Αμερική ω ένδειξη το ότι δεν μα νοιάζει το τι έγινε. Να μην το θεωρείτε δηλαδή ότι δεν μας νοιάζει η εμπιστοσύνη που πλήχθηκε η εμπιστοσύνη δική σας. Μετά από την ημέρα μου στο Βερολίνο και εδώ στις Βρυξέλλες, ακούω κάποιους που λένε ότι ανησυχούν γιατί ενδεχομένως να μην Νοιάζονται οι Αμερικανοί για τους Ευρωπαίους πλέον. Όχι. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι οι δεσμοί μας μαζί σας είναι πάρα πολύ σημαντικοί και πηγαίνουν πίσω σε βάθος χρόνου και δεν μπορούμε να τους διαρρήξουμε. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε αυτή την ρήξη στην εμπιστοσύνη. Ήρθαμε λοιπόν εδώ σήμερα. Ήταν να έρθουν και άλλα μέλη σε μια εβδομάδα εορταστική για τι ευχαριστίες, πριν τις ευχαριστίες, σε μια εβδομάδα που είπαμε στις οικογένειε μας ότι πιο σημαντικό ήταν για μας να έρθουμε εδώ να κάνουμε διάλογο μαζί μας. Γιατί είστε τόσο σημαντικοί για μας, είμαστε τόσο στενά ε, δεμένοι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το οτιδήποτε να μας χωρίσει. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με τους καλούς φίλους. Μπορεί να κάτσει κανείς μαζί τους και να τους πει την αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να κάτσουμε εδώ, να σας ακούσουμε, να τα λέτε έξω από τα δόντια και πρέπει και εμείς να σας πούμε την αλήθεια. Και πρέπει από κοινού μετά μαζί να δούμε πού θα βρούμε τον κοινό τόπο, στη μέση. Γιατί τα πρότυπα, ξέρετε, θα είναι υψηλά, ο πύχης θα τεθεί ψηλά. Και αυτό θα το θέσουμε εμείς Κανείς δεν πρόκειται να θέσει αυτά τα υψηλά πρότυπα. Εμείς θα πρέπει να θέσουμε τον πύχη λοιπόν ψηλά προκειμένου να μας ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι και όχι να δεχτούμε κάποια χαμηλά πρότυπα τα οποία ενδεχομένως να μας θέσει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ και τους τρεις σας που ήρθατε για τη συζήτηση αυτή χθες και σήμερα στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει θετική βούληση και από τις δύο πλευρές για να προκύψει η λύση. Τονίζω αυτό που μόλις είπε ο κύριος Μίξ. Το βασικό είναι να επιτύχουμε μια ε, ισορροπημένη λύση. Ξέρουμε ότι αυτά τα θέματα προστασίας δεδομένων τα αντιμετωπίζουμε από διαφορετική νομική παράδοση. Αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση γιατί δεν υπάρχουν πια σύνορα. Γιατί αυτό είναι κλασική περίπτωση όπου πρέπει να βρούμε διεθνή λύση γιατί δεν υπάρχουν πια σύνορα, δεν υπάρχει πια προστασία για τέτοια θέματα για κανέναν μόνο του. Γυρνάω προς το φίλο μου Κάλλαν. Η χώρα του ήταν το πρώτο θύμα κυβερνοεπιθέσεων. Αυτά τα θέματα λοιπόν, ιδιωτική σφαίρα, κυβερνό, εγκληματικότητα, τρομοκρατία, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με λογικό τρόπο. Αλλά είναι σαφές ότι πλήρης ασφάλεια σημαίνει πλήρης κατάρριξη της ελευθερίας. Γι' αυτό λοιπόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ελευθερία σημαίνει και κάποιος κίνδυνος. Και σε μια χώρα πλήρους ε, ασφάλειας δεν θα ήθελα να ζω. Αυτές είναι καταστάσεις που τις περιγράφει ο Huxley, ο Όουελ και άλλοι. Χαίρομαι λοιπόν για την ε, συζήτηση που είχαμε. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να σας άρεσε η συζήτηση που κάναμε εδώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη συζήτηση και εφόσον είμαστε δημοκράτες η συζήτηση μεταξύ ημών θα έχει αποτέλεσμα. Right.